Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Είναι χαρά μου να βλέπω πόσοι οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται. Εφτά λεπτά μετά την κανονική έναρξη της συνεδρίασης, πόσοι συνάδελφοι είναι εδώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με την ημερήσια διάταξή μας. Ο κύριος Μπούζεκ ζητά συγγνώμη, δεν μπορεί να έρθει. Ενδεχομένω να τον έχουμε τον απόγευμα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, οπότε θα στερηθείτε την παρουσία του. Σήμερα η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει καταρχάς τις δικές μου ανακοινώσεις. Πρώτη ανακοίνωση σήμερα το πρωί. Δεν θα γίνει καμία συνεδρίαση αύριο το πρωί. Σήμερα υπάρχει ο ε, ε, αλλά έκανε λάθος. Αύριο από τις 9 ως τις 12.30 δεν υπάρχει πρόγραμμα για την Επιτροπή μας. Δυστυχώς, εξαιτίας της παρουσίας των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε το απογευματινό μας πρόγραμμα και να το φέρουμε το πρωί. Άρα το πρωί, το πρωί δεν θα έχουμε συνεδρίαση και το απόγευμα θα συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις μας με τους εμπειρογνώμονες από τη ΣΤΟΑ. Σας ενημερώσαμε με email ότι η, η ψηφοφορία για την προφορική ε, ερώτηση ε, στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μόνο δύο σημεία στις ψηφοφορίες μας. Υπάρχει κάποια παρατήρηση για το σημερινό μας πρόγραμμα. Εάν όχι, Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, 21 Μαρτίου 2018. Υπάρχει κάποια παρατήρηση? Παρακαλώ. No message. Δεν υπάρχει. Ωραία. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Ξεκινάμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με το πρώτο θέμα, σημείο 4, πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ε, και την τροποποίηση της οδηγίας 2011-24 ΕΕ. Πρόκειται για μία έκθεση στην οποία η συγγήτρια είναι η κυρία Βίρινγκ από το Άλτε Λίβε Βίρινγκ. Έχετε τώρα το λόγο για να κάνετε την εισαγωγή. Απλά να σας ε, θυμίσω ότι μετά από 20 χρόνια εθελοντικής συνεργασίας ε, για τις ε, αξιολογήσεις των τεχνολογιών υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε πολύ ευαίσθητες περιοχές και τομείς για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός και τα ξέρω αυτά. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα είναι μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΕΜΒΗ σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Δεν βιαζόμαστε, έχουμε 30 λεπτά για αυτή τη συζήτηση. Η συγκήτρια η κυρία Βίρινγκ έχει 5 λεπτά για να παρουσιάσει τις έξοχες ιδέες της. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ εκπρόσωπε της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που είστε εδώ ως εισηγήτρια για την νομοθετική γνωμοδότηση σχετικά με τον κανονισμό HPA. Θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση στα βασικά σχόλιά μου για την πρόταση της Επιτροπής. Μετά από 20 χρόνια εθελοντικής συνεργασίας μπορώ να πω ότι χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για συνεργασία με έναν πιο συνεπή τρόπο όσον αφορά ε, στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Αυτή τη στιγμή πάνω από 58 οργανισμοί λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν αξιολογήσεις, χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες ε, υπό διαφορετικές ε, μορφές. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες είναι κατακαιρματισμένα. Θέλουμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση για τις κλινικές πτυχές αυτών των αξιολογήσεων. Ο τομέας της υγείας είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μας και αποτελεί περίπου το 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ενισχυμένη συνεργασία θα ενισχύσει και την αποτελεσματικότητα όπως ε, και το, τη σχέση κόστους-οφέλους ε, στην σχετική βιομηχανία και γενικά την ανταγωνιστικότητά μας παγκοσμίας. Γνωρίζουμε ότι οι μεθοδολογίες στην νομοθετική πρόταση δεν έχουν ακόμα καθοριστεί πλήρως. Θεωρώ ότι η ομάδα συντονισμού ως ένα κολέγιο, μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή της διαδικασίας ανάπτυξης. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, υποστηρίξει την εκτέλεση και την επιλογή των μεθοδολογιών. Ο βασικός στόχος ε, των κοινών αυτών αξιολογήσεων θα είναι να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση στη χρήση των μεθοδολογιών, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των ε, αξιολογήσεων ε, τεχνολογιών υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της συλλογής δεδομένων. Η συλλογή ποιοτικών δεδομένων είναι σημαντική για να διασφαλίσει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ικανή και συγκρίσιμη μεταξύ των κρατών μελών. Για να καταλήξω να πω ότι έχω μια σχετική ανησυχία όσον αφορά στη συμπερίληψη ιατρικών συσκευών ε, σε αυτό το νομοθετικό, σε αυτή τη νομοθετική πρόταση. Θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν ε, για την αναφορά που γίνεται σχετικά με τον κανονισμό για στις συσκευές ε, που θα τεθεί σε ισχύ το 2020. Αυτό θα είναι ε, υπό τη διαδικασία ελέγχου. Ε, χαίρομαι ε, που θα ξεκινήσει λοιπόν μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου οι παρατηρήσεις σας ακριβώς έθεσαν τον δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Ε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτά τα οποία θα βελτιστοποιήσουν ε, την εναρμόνιση. Και έχετε δίκιο, γιατί πολλοί μας κατηγορούν ότι ας πούμε κανονίζουμε παραπάνω από ότι πρέπει τις αρθρόπινες δραστηριότητες. Τώρα έχουμε τους σκιώδεις ε, εισηγητές, ο καθένας έχει Δύο λεπτά. Πρώτο το ΕΛΚ. Ο κύριος Μπουσουά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Γέρνη και τη συγχαίρω. Πολύ καλή δουλειά της, άριστη συνεργασία μας και ελπίζουμε να συνεχιστεί η συνεργασία μέχρι ό,τι ολοκληρώσουμε το θέμα. Παρά το γεγονός βέβαια ότι ίσως σε κάποια σημεία να διαφωνούμε. Έχω Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία στον τομέα υπέρ των ασθενών, των κρατών μελών και υπέρ της καινοτομίας. Εν γέννη συμφωνώ με τις ε, διατάξεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρω ότι κάποιες από τις προτάσεις ε, είναι ευαίσθητες λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής. μονούμε όμως ότι πριν από δύο δεκαετίες η ίδια συζήτηση έλαβανε χώρα με τη δημιουργία της ΕΜΑ Τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Φαρμάκων. Και τώρα η αίμα είναι επιτυχέστατο φορέα που δίνει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους Ευρωπαίου πολίτες. Εν συντομία να σχολιάσω τις προτινόμενε τροπολογίες τη ηγήτριας και ταυτόχρονα θα εκφράσω την άποψή μου. Όσον αφορά τι τροπολογίε που εξαιρούν τι ιατρικέ σχεδέ. Ε, και τις συσκευές ε, σε, σε εργαστήρια έχω κάποιες αμφιβολίες. Η τεχνολογία αξιολόγηση, η τεχνολογική των ιατρικών συσκευών ε, δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα εν συγκρίση με τα φάρμακα. Αλλά είναι περιορισμένο το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού σε συσκευές υψηλού κινδύνου ταξινομίες 2β, 3 και 4 δέλτα και εκεί υπάρχει έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό περιατρικών συσκευών. Και το άρθρο 5.2 τη πρότασης καθορίζει καθηγητέ γραμμές του πότε λαμβάνει η χώρα με τη ταξιολόγηση. Και πιστεύω ότι οι διατάξεις δεν θα επιβαρύνουν τους αρμοδίους που κατασκευάζουν συσκευές, θα είναι υπέρ των ασθενών παρόμοιες, ε, ε, παρόμοια έλεγχοι ε, ήδη εφαρμόζονται. Το πεδίο εφαρμογή είναι περιορισμένο, ευρύ 2006 ευρύ το χρονικό περιθώριο για τις ιατρικές συσκευές του 2020 και 2022 για τη διαγνωστική in vitro. Όσον αφορά τροπολογία 18 που μπορεί η αρμόδια ομάδα να επιληφθεί και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς σαν Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί, να δώσουμε την ελευθερία στους εμπειρογνώμους που προσωπούν τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν τους δικούς τους κανόνες, τους διαδικαστικούς Καλύτερα να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω σε αυτή τι αρμοδιότητες μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων για του διαδικαστικού κανόνε Και ζητώ από την εξηγήτρια να εξηγήσει κάπω κάτι, παρόλο που το συζητήσαμε. Πολλοί συνάδελφοι και συνεργάτε μου δεν κατάλαβαν πλήρω αυτό που θέλω να ζητήσω. Την τροπολογία 22, κυρίω το δεύτερο τμήμα τη 22, της παραγράφου 2 και τώρα είμαι υπέρ της καινοτομίας και πιστεύω ότι διαδικαστικές και μεθοδολογικές ε, ε, διατάξεις για την αξιολόγηση και διαδικασίες για κοινή επιστημονική διαβούλευση θα πρέπει να επικαιροποιούνται συνέχεια ώστε να προσαρμόζονται στις επιστημονικές εξελίξεις και να υπάρχει και παρκής ε, ευελιξία ούτως ώστε να γίνεται παρκής αξιολόγηση των τεχνολογιών της, του τομέα της υγείας. Αυτά και ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ξεπεράσατε κατά 1,5 λεπτό το χρόνο σας, όμως η ιδέα σας είναι πολύτιμη. Πάντα πρέπει να ακολουθούμε το ρυθμό της προόδου. Διαφορετικά κάπου θα κολλήσουμε. Θα σταματήσουμε και θα παρακολουθούμε τους άλλους που θα προχωρούν. S&D τώρα. Ο Πόπα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Χαιρετίζω από την πλευρά μου την πρωτοβουλία της Επιτροπής ε, για μια καλύτερη βάση αυτές τις συσκευές και τις τεχνολογίες. Ε, μιλάμε για συσκευές ιατρικές ε, που στην ουσία αφορούν ασθενείς ε, και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι ιατρικές συσκευές θα πρέπει να αξιολογούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα διότι όπως είπα είναι σημαντικά και για τους ασθενείς αλλά και για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι επίσης σημαντικό τα δεδομένα που συλλέγω ε, από τα κράτη-μέλη να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους ε, και να υπάρχει μια διαφάνεια σε αυτή την διαδικασία γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους μητρώα δεδομένων. Η διαλειτουργικότητα επίσης, διασυνδεσιμότητα είναι ε, μια απέτηση. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μια τυποποίηση των μεθοδολογιών οποία, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά συγκρίσιμες. Θέλουμε να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να εισαγάγουμε μία βασική συνεργασία στον τομέα αυτό, ε, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τους πόρους που έχουν διαθέσιμους. Θεωρώ επίσης ότι η προστασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ε, την εμπιστευτικότητα. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για την προστασία των ε, ασθενών. Επίσης, ε, τα ευρήματα για σπάνιες ασθένειες ε, θα πρέπει να συγκρίνονται για να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση. Επίσης, ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα να εισαγάγουμε ένα κεφάλαιο σχετικά με τις συγκριτικές μελέτες ε, το οποίο θα μιλά για τις ε, μεθόδους ε, θεραπείας. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοια δεδομένα για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις τεχνολογίες υγείας. Έτσι θα έχουμε πιο αποτελεσματική εργασία και θα έχουμε καλύτερη αξιολόγηση της θεραπευτικής αξίας αυτών των συσκευών. Ευχαριστώ. Well, Σας ευχαριστώ πολύ. Το σχόλιο σας για την προστασία δεδομένων είναι πολύτιμο. Όμως η υπερβολική ρύθμιση του τομέα θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για την ανάπτυξη κάποιων ιατρικών ε, συσκευών. Διότι υπάρχει τεράστιο φάσμα δυνατοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων. Και κάπου κάπου μπορεί να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ προστασίας δεδομένων και περαιτέρω ανάπτυξη ε, τέτοιων συσκευών. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί κανονισμοί. Άλλος σκιώδης, παρίσταται άλλος σκιώδης, ο οποίος θέλει να, να ακουστεί η φωνή του στη συζήτηση. Αν δεν υπάρχει, άλλα μέλη. Έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον ένα λεπτό ο καθένας αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι σχετικά με αυτό το θέμα αν δεν θέλει να μιλήσει κανείς θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε χρόνο μέχρι και τρίλεπτο για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Αμπελάς έχει το λόγο ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε στη συζήτηση και ευχαριστώ και την εισηγήτρια, την κυρία Βιέρνικ, για τη γενική υποστήριξη που μας έδωσε στην έκθεση και που μας υπενθύμησε ότι αυτό το έργο δεν ξεκινά τώρα με αυτή την πρόταση, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια αυτή η συνεργασία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρήσαμε ότι σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να αυξηθούν οι δεσμεύσεις ε, στον τομέα αυτό. Και αναφέρθηκαν σημαντικές πτυχές στη συζήτηση. Πρέπει να αυξηθεί η προσέγγιση βάση στοιχείων και να προωθηθεί καινοτομία. Αυτό προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε στην πρόταση. Κάποια σχόλια έχω, κυρίως για τις ιατρικές συσκευές και τα σχετικά σχόλια. Προετοιμάζοντας την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε προσεκτικότατα τις εκφραστήσεις ανησυχίες του τομέα που κατασκευάζει τις συσκευές. Έχουμε επίγνωση των ανησυχιών τους. Προσπαθήσαμε παντιοτρόπως να λάβουμε υπόψη στην πρότασή μας ανησυχίες. Αν δούμε το πεδίο που καλύπτεται, όπως αναφέρθηκε από το συνάδελφο Μπουσόη, το πεδίο εφαρμογή που καλύπτεται στις συσκευές είναι πολύ περιορισμένο στην πρόταση. Μόνο στις ιατρικές συσκευές επικεντρωνόμαστε όπου υπάρχει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία. Δηλαδή, στις συσκευές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τις ανάγκες των κρατών μελών εστιαζόμεθα μόνο επ' αυτών των ιατρικών συσκευών που ήδη έχουν περάσει από διαδικασία ελέγχου έχει ήδη τοποθετηθεί το πάνελ των εμπειρογνωμόνων επ' αυτών και πέραν αυτού πρέπει να επιλεγούν από την ομάδα συντονισμού που αποτελείται από από μέλη. Οπότε το ε, πεδίο υποχρεωτική εφαρμογή είναι περιορισμένο έτσι ιατρικέ συσκευέ. Επιτρέπει μεγάλη ευελιξία για την ομάδα συντονισμού να αποφασίζει σε ποια ιατρική συσκευή θα ήθελα να υπάρξει συνεργασία. Πέραν αυτού παρέχεται και δυνατότητα και προθυμία υπάρχει για συνεργασία σε άλλους τομείς. Και αυτό όμω επιθελοντική βάσεω. Μετά αν δούμε το χρονικό ζήτημα στην πρότασή μας εξασφαλίσαμε ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν αλληλοκαλύπτονται. Η πρότασή μας, εάν υιοθετηθεί, η πρώτη προθεσμία εφαρμογή αν όλα πάνε καλά, της προτάσεως θα είναι το 2023, λίγο πολύ, και, και ο κανονισμός ιατρικέ συσκευές ήδη θα έχει εφαρμοστεί τότε. Άρα δεν διαβλέπουμε πρόβλημα όσον αφορά επικάλυψη πλευρά χρονοδιαγραμμάτων, αλλά είναι θέμα να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις δύο διαδικασίες, να χρησιμοποιηθεί κάποια τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται στον τομέα των ιατρικών συσκευών και για το κοινό κλινικό αυτό έργο. Τρίτο που ήθελα να αναφέρω αφορά τις ιατρικές συσκευές και αφορά την ευελιξία που προβλέπεται από την πρόταση. Παραδεχόμαστε ότι ο χρονισμός για την κοινή κλινική αξιολόγηση μπορεί να λάβει χώρα αργότερα από ό,τι προβλέπεται για τα ιατρικά προϊόντα μετά την διάθεση στην αγορά και η πρόταση αναγνωρίζει επίσης τις ιδιαιτερότητες των ιατρικών συσκευών και του σχετικού τομέα και επιτρέπεται μέσω κατεξιδότησης συμπράξεως να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα και διάφορες ομάδες και επιτροπές υπό διάφορες συνθέσεις να συναντώνται όταν μιλάμε για τα ιατρικά προϊόντα, για τα φαρμακευτικά προϊόντα ή τις ιατρικές συσκευές. Έτσι προσεγγίσαμε το θέμα. Κατά κλείδι πιστεύω ότι υπάρχει μικρό πεδίο για τι ιατρικέ συσκευέ. Λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίε που εκφράστησαν από το τομέα και επιτρέπουμε δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας αν υπάρχει ενδιαφέρον αυτά και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τα όσα εσείς υπογραμμίσατε είναι πολύ σημαντικά δεν μπορούμε εμείς να εντάξουμε ιατρικές συσκευέ οι οποίες είναι ενδεχομένως επικίνδυνες για τους ασθενείς. Η κυρία Βίριν για να κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια ε, τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το φάκελο αυτό. Η συνεργασία μεταξύ μας ήταν πάρα πολύ καλή και αυτό το οποίο εκτιμήσα ιδιαίτερα ήταν η ευελιξία με την οποία εργάστηκαν. Είμαι σίγουρη πως όλοι μαζί θα καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ και εγώ. κυρία Καβεσόν Ρουίς ε, ε, εμπνεύστηκε από την ε, παρέμβασή σας και ζητά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ζήτησα το λόγο προφανώς δεν με είχατε δει. Φαντάζομαι ότι η συγγήτρια αν χρειαστεί θα μου απαντήσει. Πιστεύω πως η πρόταση είναι σημαντική, δίνει προσθέμενη αξία, δίνει ευρωπαϊκή αξία και είναι ε, μία από τις ε, προσπάθειες που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε την εκτιμώ ιδιαίτερα θετικά. Είναι σημαντικό να δούμε και την πλευρά της βιομηχανίας αλλά και της έρευνας. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει καλύτερο η εσωτερική αγορά ε, και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις αρμοδιότητες της δική μας Επιτροπής, αλλά να δούμε και το τι χρειάζεται να κάνετε τη στιγμή αξιολόγηση στο κάθε κράτος μέλος για να δούμε ε, πώς θα λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτή τη στιγμή ε, οι εταιρείε δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα παρόλο που κυκλοφορούν τα προϊόντα τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές δεν έχουμε αρκετά τεκμήρια για να κάνουμε την κατάλληλη αξιολόγηση. Πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και κάτι ακόμα γιατί πολύ συχνά έχουμε υψηλές τιμές ε, γιατί δεν έχουμε τις απαραίτητες ε, κλινικές ή ιατρικές πληροφορίες. Άρα λοιπόν χρειάζεται η ποιότητα της έρευνας να βελτιωθεί και να έχουμε περισσότερα τεκμήρια και αποδεικτικά στοιχεία και δοκιμές για να είναι περισσότερος ο ανταγωνισμός και να είναι πιο ποιοτικά ε, τα προϊόντα που μπαίνουν στην αγορά. Θα ήθελα να εστιάσω σε ένα μάλλον επίμαχο που είναι αυτό των ιατρικών συσκευών. Πιστεύω πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο τολμηρή ε, και θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε την κατάλληλη ε, αξιολόγηση αυτών των συσκευών και ε, ε, ε, και να έχουμε καλύτερη ποιότητα έρευνας με μια σταδιακή αύξηση των απαιτήσεων από κάθε κράτος μέλος γιατί νομίζω όλοι ζητάνε αυτή την απαραίτητη συνεργασία έτσι ώστε τα στοιχεία και τα, τα, δεδομένα να λαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο υπόψη από όλους. 20 τέτοιοι οργανισμοί υπάρχουν σήμερα γίνονται λοιπόν 20 διαφορετικές αξιολογήσεις, όπως γίνεται και για τα φάρμακα. Καλό είναι να έχουμε λοιπόν περισσότερο διάλογο, να βοηθηθούμε και να έχουμε περισσότερη συγκρισιμότητα στον κλάδο. Ο κανονισμός οδηγία για τις ιατρικές συσκευές που θα, μπεις, θα τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να εστιάζει κυρίως ε, στην ασφάλεια. Αλλά δεν έχουμε καμία εξασφάλιση πως θα είναι και αποτελεσματικά και αποδοτικά. Έχουμε και ηθικά διλήμματα. Όταν εγκρίνουμε ένα φάρμακο, μια ιατρική συσκευή, είναι ένα υγειονομικό προϊόν που πρέπει να είναι ασφαλές, αλλά θα πρέπει να είναι και αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν είναι ε, καλή η πορεία που ακολουθεί αυτό το κείμενο, ε, για το θέμα της ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να ε, βελτιωθεί ε, για το κομμάτι που έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα αυτών. Και νομίζω πως για τις ιατρικές συσκευές, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αξιολογούμε όχι μόνο αυτές που είναι υψηλού κινδύνου, αλλά όποια αποτελούν καινοτομία και μπορεί να έχουν συνέπειες για τη δημόσια υγεία ή που μπορεί να έχουν κάποιες δημοσιονομικές επιπτώσεις του προπολογισμού των ε, κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω οι αξιοσημείωτες ιδέε σα να είναι χρήσιμες στη συνάδελφο, την κυρία Βίρινγκ. Well, uh, I think we have to mention... Λοιπόν, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 23 Μαΐου μεσημέρι, δηλαδή στις 12. Και θα ψηφίσουμε στην Ήτρε στις 9 Ιουλίου του 2018 στην έμβη η ψηφοφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί Δηλαδή μετά τη δική μας ψηφοφορία στην Ίτερ θα περάσει και από την αρμόδια επιτροπή που είναι η ΕΝΒΗ και θα πάει στην Ολομέλεια σύμφωνα με τις προβλέψεις μας 1η Οκτωβρίου φέτος. So, we can conclude by these remarks. Λοιπόν, με αυτά τα σχόλια μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο και μετά να περάσουμε στην απόφαση για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τροπολογίας στο Μνημόνιο Συνεργασίας ΝΑΤ 19406 μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο πρώτος σκιώδης είναι έτοιμος. Έχω δει και την κυρία Κέλλη και τον κύριο Κέλλη, με συγχωρείτε, ε, και Νομίζω ότι και άλλοι θα θελήσουν να πάρουν το λόγο να σχολιάσουν. Να πω και εγώ δύο λόγια. Το πρώτο, το, η πρώτη αυτή τροποποίηση ε, ε, διαπραγματεύτηκε ε, μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας για τις αερομεταφορές των Ευρω... Ε, Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με υπογραφή στη 13 12 του 2017. Το 60% των αερομεταφορών ε, γίνεται με μεταφορικές εταιρείες αεροπορικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, των ΗΠΑ και σύμφωνα με τα 102 και 118 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να εγκρίνει αυτή την ανανέωση την οποία μόλις σας περιέγραψα. Σας ενημερώνω πως έχουμε στη διάθεσή μας χρόνο μέχρι τις 10. Εκεί θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ πολύ μην το ξεχνάτε. Δίνω τώρα το λόγο στον ε, εισηγητή, τον κύριο Πάξα, για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Έχετε τρία λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε το λόγο. Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας ε, πρέπει να το σχολιάσω με τρόπο στοχευμένο, με τρόπο σύντομο και με τρόπο συγκεκριμένο είναι ένα μνημόνιο συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο από το 2011 και μετά είναι σε ισχύ. Έκτοτε, τα αποτελέσματα είναι αυτά και πρέπει να σας πω πως η έρευνα και η τεχνολογία στην διαχείριση εναέρειας ε, κυκλοφορίας έχει λάβει σάρκα και οστά με τα διάφορα ε, project ε, που είναι το Next Gen για παράδειγμα και το πρόγραμμα για την ε, εναέρια κυκλοφορία και πρέπει να σας πω πως η συμφωνία θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του μνημονίου για να καλύπτει όλες τις φάσεις του εξυγχρονισμού της εναέριας κυκλοφορίας και σε αυτό ε, θα συμπεριλάβουμε και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερο το πεδίο εφαρμογής ε, συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων οργάνων ε, των δύο μερών και για να ληφθούν όντω υπόψη και όλες οι εξελίξεις στην τεχνολογία πολιτικής αεροπορίας. Η προτινόμενη απόφαση ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι συμπίπτει απόλυτα και με τους πολιτικούς στόχους που έχουμε ε, τοποθετήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Νομίζω ότι τώρα ήρθε ο... η στιγμή να δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Βλέπω τον κύριο Κέλλη, είναι έτοιμος. Κάθε σκιώδης έχει στη διάθεσή του δύο λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης σε αυτό το στάδιο το χαιρετίζουμε. Διότι συνεχώς συζητάμε για την έλλειψη συνεργασίας και την απόκληση των δύο μερών μεταξύ τους. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Φυσικά πρέπει αυτά τα θέματα να τα δούμε μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε και τα όσα κάναμε ως τώρα, σε μακρόπνο επίπεδο. Αυτή η συνεργασία, το μνημόνιο συνεργασίας είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδα μεταφορών. Επίσης, ε, η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ουρανών είναι ύψης της σημασίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή. Να συνεχίσουμε τη συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν οι ανοιχτοί ουρανοί, το Open Skies. Να υπάρχει μια εγγύηση για την ασφάλεια των επιβατών και να υφίσταται η βέλτιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ της δικής μας πλευράς εδώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό επιθυμούν όλοι. Και ο εισηγητής, ο κύριος Πάξας, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι αυτό θα συνεχιστεί. Θετικά όλα αυτά λοιπόν και συνυπογράφω. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Είναι κάποιος που θέλει να εκφράσει κάποια άποψη από την πλευρά των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Όχι. Ο κύριος Τσέσακ τότε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Παρόλο που θα συζητάμε το ε, θέμα στο επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, νομίζω ότι στο θέμα της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ η συνεργασία στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω σε τέτοια παραδείγματα. Το μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΕ όσον αφορά στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας το 2011 είχε να κάνει με τα συστήματα διαχείρισης και κυκλοφορίας, τα λεγόμενα ATMs αλλά και την έρευνα και ανάπτυξη μετά από ένα συγκεκριμένο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης ε, που μας έφερε πολλά ωφέλη σε επίπεδο παγκόσμιας διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ, ΕΕ, τώρα ε, έχουμε το επόμενο λογικό στάδιο της στρατηγικής. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Συμβουλίου να ανανεώσει και να επεκτείνει το μνημόνιο σε ένα νέο στάδιο εφαρμογής. Ελπίζουμε ότι η εφαρμογή των συστημάτων ATM θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την εσωτερική μας αγορά επίσης, ότι θα ευνοήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας μας. Εκ μέρου της πολιτικής μας ομάδας ε, θα ήθελα να πω ότι επιβεβαιώνουμε την προσέγγιση του εισηγητή και υποστηρίζουμε την επέκταση αυτού του πρωτοκόλου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μια ιδανική κατάσταση. Όλοι συμφωνούμε με τον εισηγητή. Είναι κάποιος που θα ήθελε να εκφράσει κάποιες άλλες ιδέες για αυτό το θέμα, τις ιδέες του για αυτό το θέμα. Όχι. Κανείς δεν εκδηλώνει τέτοια επιθυμία και από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει και κάποιος από την Επιτροπή. Α, όχι, η κυρία Βιρνίκ. Έχετε κάποια ερώτηση για την Επιτροπή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μας την απαντήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Μάισνερ, που είναι η σκιώδης για το, α, εκ μέρους του Άλτε, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή. Θεωρεί ότι στον τομέα της ε, πολιτικής αεροπορίας είναι πολύ σημαντικό να ευνοήσουμε τα διεθνή σάνταρ, γιατί αυτό προωθεί τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την επέκταση αυτού του μνημονίου συνεργασίας. Αυτό θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΙΠΑ να συνεργαστούν ακόμα περαιτέρω για τον εξυγχρονισμό των συστημάτων διαχείρισης εναέρεια κυκλοφορίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Από όσο γνωρίζω, η κυρία Μάισνερ γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα γιατί έχουμε συνεργαστεί στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχουμε ήδη θέσει κάποια στάνταρ που ισχύουν για όλο τον κόσμο. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη μόλις έφτασε και θα ήθελα να κάνει κάποιο σχόλιο για αυτό το θέμα από ό,τι βλέπω. Ναι, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Μιλάμε για τη συνεργασία μεταξύ ΕΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης και κυκλοφορία. Όπως ε, υπόθηκε ήδη, η τροποποίηση του μνημονίου για να προχωρήσουμε από την έρευνα και την ανάπτυξη στην εφαρμογή και εκτέλεση ε, θα βοηθήσει την συνεργασία μας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Ε, να σας ε, θυμίσω ότι οι αεροπορικές μεταφορές έχουν ραγδαία αύξηση 7,8 δις επιβάτες είχαμε το 2016 και αναμένουμε διπλασιασμό. Υπάρχουν λοιπόν πολλαπλές προκλήσεις. Το ίδιο το θέμα ε, είναι με γεμάτο προκλήσεις γιατί πρέπει καταρχάς να διασφαλίσουμε ότι θα προστατέψουμε από την υπερθέρμανση του πλανήτη, να έχουμε βελτίωση των τεχνολογιών, αλλά θέλουμε και να ενισχύσουμε και το ρόλο των βιοκαυσίμων στην αεροπλοεία. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία θα μας βοηθήσει σε αυτό το τομέα για τα βιοκαύσιμα ε, έχουμε ήδη ε, καταθέσει το 3 και το 1 και ελπίζουμε ότι θα μείνει στον τριμερή διάλογο. Επίσης θέλουμε καλύτερη ασφάλεια, ειδικά στα πιο ε, ας πούμε πολυπληθή και αποσχολημένα αεροδρόμια του κόσμου. Για να μην λέω πολλά, νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε περισσότερες, περισσότερη συνεργασία μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζω τον εισηγητή και τη σύστασή του. Ευχαριστούμε πολύ για τις αξιόλογες παρατηρήσεις σας. Νομίζω ότι η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Ως τώρα η πολιτική αεροπορία έχει ε, και όλα αυτά τα θέματα τα περιβαλλοντικά που είπαμε. Ε, νομίζω ότι ε, βέβαια ήδη έχουν γίνει κάποια πράγματα σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, αλλά περιμένουμε και άλλα. Τώρα έχουμε λοιπόν τον λόγο, τώρα έχουμε λοιπόν τον εισηγητή. Ο εισηγητής μας έχει το λόγο. Έχει. Κύριε Πάξας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι ευγνώμων που στηρίζετε τη θέση μου να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ στον τομέα της ε, έρευνας και ανάπτυξης για την διαχείριση της και κυκλοφορίας είναι πολύ σημαντική και χαιρετίζω τα σχόλια και την υποστήριξή σας. Ελπίζω όλα αυτά να συμπεριληφθούν στο κείμενο και να τα υποστηρίξετε και με την ψήφο σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για αυτά τα σχόλιά σας. 9 και 47. 13 λεπτά στη διάθεσή μας. Μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. Καταληκτικά σχόλια. Ο χρονισμός. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 23 Μαΐου. Το μεσημέρι στις 12. Ψηφοφορία στην Ήτρε 19 Ιουνίου του 2018. Στην Ολομέλεια ψηφοφορία αναμένεται το Σεπτέμβριο ενεστώτος έτους. Ευχαριστώ. Σύντομο διάλειμμα μέχρι τις 10 που θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Να πάτε να φρεσκαριστείτε κάπως.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Α, σου έρθει η dear colleagues, it's 10 o'clock. Αγαπητοί συνάδελφοι, ώρα 10. To ask you to... Καθίστε παρακαλώ. According to the program, we have to start the first... Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο σημείο της ψηφοφορίας μας. Παρακαλώ, πιάστε τις κάρτες σας, όχι με τη διεύθυνσή σας, αλλά ψηφοφορίας. Παρακαλούμε να συσαχθούν οι κάρτες στο ηλεκτρονικό σας μηχάνημα. Πρέπει να διερευνήσουμε τον αριθμό των παρόντων από κάθε ομάδα. Κυρία Τόγια ψάχνει την κάρτα της. Να σας δανείσω καμιά καρτούλα. Ποιος έχει πάρει την κάρτα της κυρίας Τόγια. δεν μας προσέχουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας όπως πρέπει. Λοιπόν, τόσες κάρτες υπάρχουν. Okay, uh, well, let's, let's start. Ας ξεκινήσουμε. Να κάνουμε μια δοκιμή, να ξέρουμε πώς είναι παρόντες από κάθε ομάδα. Παρακαλώ, πατήστε ναι. Ποιος είναι πράγματι παρόν, πατήστε το ναι. Ξεκινάει η ψηφοφορία, η δοκιμαστική. Did everyone vote? Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Πρόεδρε, Ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω την κάρτα μου, αλλά είμαι παρόν. Να προσθεθεί η μου στην ψήφο του ECR. Θα μετρήσουμε δύο συν από κάθε ομάδα. Τρεις. Ωραία. Λειτουργεί στην συγκεκριμένη περίπτωση ακόμα και το ΕΛΚ δεν έχει παραπάνω μέλος όπως συνήθως από ό,τι θυμάμαι. Ξεκινάμε λοιπόν. Μία ψηφοφορία επί προφορικής ερωτήσεως για την τεχνολογία των αρχείων και των blockchains ε, δημιουργώντας ένα κλίμα η κυρία Εύα Τελική ψηφοφορία όσον αφορά την προφορική ερώτηση. Ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ, μάλλον άρχεται η ψηφοφορία, λέει ο Πέρες. 55 συν η κυρία Τόγια που είναι υπέρ. Ας ελπίσουμε να βρει βοηθό σας την κάρτα σας. Πρόεδρε, ποια είναι η μοναδική ψήφος η αρνητική παρακαλώ. Θα, θα ξέρουμε ποιος ψήφισε κατά. Αστιάκι ήταν λέει ο κ. Μπουτικόφερ. Θα δημοσιευτεί λέει ο πρόεδρος. Σας αρκεί αυτό, σας καλύπτει. Πάμε παρακάτω. Πρόταση ψηφίσματος. Ησυχία παρακαλώ. Με την λογική αναφορά 10. Τροπολογία 1. Θέση εισηγήτριας υπέρ. ποιο είναι υπέρ. Κατά. άποχέ Δεχτή. Συμβιβαστική 1. Εταιρική σκέψη α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά άποχες δεκτή συμβαστική 3 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή σημαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτωτα. Είσαστε υπέρ. Μάλιστα αποφασιστική ψήφος. δεκτών. Τροπολογία 22 δεκτή. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Άποχες ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 24. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 29 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 30 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 31 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 32 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 41 εάν εγκριθεί καταπίπτει η τροπολογία 42 υπέρ τη 41 κατά άποχες εγκρίνεται οπότε 42 καταπίπτει τροπολογία 43 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 44 υπέρ κατά Αποχές. Έλεγχος. Τροπολογία 44. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ που περισσεύει. Αυτό μου αυτό μου λείπε. Αυτό μου ξέφευγε πάντα. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά άποχες έλεγχος. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 55 ονομαστική. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. δεκτή. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεχτεί. Σημαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68 αν εγκριθεί καταπίπτει η 69. Υπέρ λοιπόν της 68 παρακαλώ. Κατά. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η, η τροπολογία 69. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 Είπε. κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβιβασ... Μάλλον, τροπολογία 93 Είπε. κατά άποχες απορρίπτωτα. Τροπολογία 94 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Εντάξει, αν το χρειάζεστε και το ζητάτε, αν το κάνουμε. Τροπολογία 98, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάμε. Τέλος ψηφοφορίας. Ξεκάθαρο. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 107 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 116 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Δεν είναι ξεκάθαρη κατάσταση για την 116 ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνοντα. 117 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε για την 117 ηλεκτρονικό έλεγχος που άρχεται. Ξεκινάμε λοιπόν. Πέρας. Σαφής η αποδοχή της τοπολογίας. 118. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 128 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 129 υπέρ κατά Αποχές. Έλεγχος για την 129. Άρχεται. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Αποφασιστική διαφορά. Παρά το γεγονός δεν ήταν ξεκάθαρο οπτικά. Τροπολογία 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 132 εάν εγκριθεί αυτή οι 133 και 134 καταπίπτουν οπότε 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 αν εγκριθεί πίπτη 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 133 πέρας ένα μέλος του ΕΛΚ περισσεύει μπορεί να διεθώσετε παρακαλώ Καλώς. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. 134 καταπίπτει, 135 υπέρ, κατά άποχες, έλεγχος. 135 άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος, πέρας, εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 137 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 138 αν εγκριθεί κατά πίπτη 139 138 λοιπόν υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 138 έλεγχος για την 138 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 139 κατά πίπτη οπότε πάμε στην 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά Αποχές. Έλεγχος. 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 142. Αν εγκριθεί κατά πίπτη 143. Ποιος είναι υπέρ της 142. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 143 καταπίπτει, 144 εάν εγκριθεί καταπίπτει 145. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145, 145 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 145. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Η ίδια διαφορά φαίνεται και εδώ. Δεκτή. 147 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 147 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. 148. Πέρας για την 148. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 152. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 159 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 159 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 160 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 161 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 162 αν εγκριθεί καταπίπτει 164. Λοιπόν, 162 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 163, αν εγκριθεί πίπτη τροπολογία 164, οπότε τροπολογία 163 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 164 κατά πίπτη 165 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 166 πίπτη, Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182, αν εγκριθεί καταπίπτει 183, είναι υπέρ της 182, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 184 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 αν εγκριθεί κατά πίπτη τροπολογία 187 υπέρ της 186 κατά αποχές εγκρίνεται 187 κατά πίπτη 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 190 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 191 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος ως ετροποποιήθη ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται. Πέρας. 52 υπέρ, μία ψήφος κατά, έξι εποχές, μεγάλη διαφορά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Καηλή. Υπέροχα. Well, the next Η επόμενη ψηφοφορία είναι για μία προφορική ερώτηση που έχει να κάνει με την έκθεση Μάρκους Πίπερ. Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν και θα ξεκινήσουμε υπέρ. Λίγη. 47-10, μεγάλη πλειοψηφία, σας συγχαίρω. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο ψήφισμα που δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπέρ συμβιβαστική 1 κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 23, συγγνώμη, η τροπολογία 25 αν εγκριθεί καταπίπτουν 23 και 24. Υπέρ. Στην 25 πάντα Κατά. Απορρίπτεται. 24. Α, για την 25. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. 24. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 23, τροπολογία 26. Εάν εγκριθεί, καταπίπτει 27. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27. Για την 26. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Πάμε στην 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ξεκάθαρα. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Στη σελίδα 4 είμαστε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ. Κυρία Τόια είναι υπέρ λοιπόν. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την 79. 79. άρχιτη ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 82. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 Δύο σελίδες παρακάτω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Στη συμβιβαστική τροπολογία μόνο 8. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Λοιπόν, απορρίπτεται. Θα ακολουθήσουν λοιπόν η 91 και 92 μαζί. Ε, later, my dear. So, amendments number... Περνάμε λοιπόν στην 91 και 92 που θα τις δούμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Την 96. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ξεκινάει. Λήξη. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Είμαστε στην 99. Ελέγχουμε την 99. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 98. Γιατί επειδή εγκρίθηκε η 99 καταπίπτουν οι 97 και 101. 98 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Άποχες, απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Άποχες, απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Άποχες, εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά εδώ λοιπόν να τη δούμε ηλεκτρονικά την 108 ξεκινάει η ψηφοφορία λήξη απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά εγκρίνεται 113, 114, 115 και 117 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα την 111. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την 111. Άρχεται η ψηφοφορία 111. Λήξη. Εγκρίνεται. 105, 108, 112, 113, 116. Εγκρίνεται. 14 και 15 καταπίπτουν, ψηφίζουμε την 106. Από, αν εγκριθεί, καταπίπτουν και 107. Υπέρ. Στην 106 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. 106. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ την 110 άρχεται πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ τη συμβιβαστική υπαρθμόν 9 ε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Κατεβαίνουμε κάτω μία σελίδα. Είμαστε συμβιστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην 141, στο δεύτερο τμήμα, το κείμενο που λέει «Therefore urges the Commission 25% από τον ορισμό των μικρομεσαίων». Οπότε το κομμάτι αυτό, το δεύτερο τμήμα της 141, θα ψηφιστεί τώρα. Υπέρ. Κατά. Θα το δούμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 142. Για την 142 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκεί τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. C. Συμβιβαστική C. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Εάν εγκριθεί, καταπίπτουν 14 και 15. Οπότε, 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Εάν εγκριθεί, έχει καταπέσει ήδη 13, εν πάση 14, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. 14. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 18 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται Τελική λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο. Ε, αρχίζει η ψηφοφορία, ανοίγει. Λίγη. Ξεκάθαρα γίνεται δεκτή και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρασε λοιπόν εδώ τελείωσε το όλο θέαμα κυρία Τόια, εγκρίθηκε στη δεύτερη ψηφοφορία. So now it's time to make a short... Οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Μπορείτε να ανταλλάξετε τις ε, ξέρετες απόψεις σας με τους συναδέλφους σας και μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε σε δύο λεπτά. Και 50 δηλαδή. Δύο λεπτά. job, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ζητήσω να ολοκληρώσετε τις ε, προσωπικές σας συζητήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας. Το επόμενο θέμα, εάν δεν σας ενοχλώ αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Μην ενοχλείστε, απλώς βγείτε έξω και μπορείτε να συζητήσετε όσο θέλετε. Βασικά πρέπει να συζητήσουμε την επέκταση της Συμφωνίας για την Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρόκειται για εξέταση του σχεδίου έκθεσης εισηγητής Ρολάντας Πάξας. Είναι μια διαδικασία συνένεσης για να επεκτείνουμε την υφιστάμενη συνεργασία σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια τέταρτη επέκταση της συμφωνίας και ο σκοπός της οποίας είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις ε, συνεργασίες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ε, έρευνα και ανάπτυξη ε, επιστήμης και τεχνολογίας. Η υφιστάμενη συμφωνία λήγει τον Οκτώβρη. Έτσι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το θέμα σε μια επίγουσα διαδικασία τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε συγκεκριμένο χρόνο. τουλάχιστον 10 λεπτά. Κύριε Πάξας, θέλετε να μας παρουσιάσετε το σχέδιο της έκθεσης. Έχετε το λόγο. Ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όντως η συνεργασία, η συμφωνία συνεργασίας σε τομείς επιστήμης και τεχνολογίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ ισχύει ήδη από το 1998 ε, με διάφορες επεκτάσεις. Τον Οκτώβριο του 2018 λύγει η τρίτη επέκταση. Ε, η πρώτη ήταν ε, το 2003 μετά το 2008 και μετά το 2013. Ε, μπορούν οι περιφέρειές μας και τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές. Έχουμε δει πολύ ε, καινοτομία και μεγάλες αλλαγές βάση αυτού. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η ΕΠΑ είναι πολύ σημαντικός ε, εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα της καινοτομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών σε αυτόν τον τομέα. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό η συμφωνία σε αυτόν τον τομέα να επεκταθεί για άλλα πέντε χρόνια. Αυτό θα διασφαλίσει την προώθηση στρατηγικών συμπράξεων και θα ενισχύσει την αμοιβαία υποφελή συνεργασία προωθώντας ε, ευνοϊκές συνθήκες ε, για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θεσμών εργασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Θέλω να πω ότι υποστηρίζω αυτή την ε, πρόταση. Ευχαριστούμε κύριε Πάξας. Τώρα ήρθε η ώρα οι σκιώδεις να εκφράσουν τις απόψεις τους. Δύο λεπτά ο καθένας. Ελκ. Κανείς. Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες, κανεί. ECR, ο κύριο Τσέσακ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο δεύτερη φορά όσον αφορά το κεντρική σημασία ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΕ αυτή τη φορά για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια πολύ ενεργή τρίτη χώρα του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Έχουμε πολλούς επιστήμονες που συνεργάζονται. Έχουμε ε, κοινέ πατέντες, δημοσιεύσεις, κοινά προγράμματα, κοινή έρευνα. Και γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Συμβουλίου για την επέκταση της συμφωνίας, διότι η Ευρώπη θα πρέπει γρήγορα να αναλάβει πρωτοβουλία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες ψηφιακές προκλήσεις για την οικονομία μας. Είναι λοιπόν λογικό να ενισχυθεί η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού όπως ανέφερε και ο εισηγητής. Η συμφωνία επίσης είναι ένας τρόπος να εργαστούμε επί μίας ολοκληρωμένης ε, στρατηγικής ε, που θα ενισχύσει μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση και εσωτερικοποίηση της ε, καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επέκταση τη συμφωνίας ε, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν πρόσβαση σε επιστημονικές ε, και εξειδικευμένες γνώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχουμε και περισσότερα προγράμματα, περισσότερες ανταλλαγές σε επίπεδο γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας. Αγαπητέ εισηγητά, υποστηρίζουμε τη θέση σας. Πρόκειται για μια εκτεταμένη έκθεση, ένα σχέδιο έκθεση. Ε, ιδιαίτερα εκτεταμένο, ε, εξαντλεί όλα τα θέματα, δεν θα υπάρξουν πρωτοπολογίε από εμά. Ωραία. Ο εκπρόσωπος του Άλντε, ο Πρόεδρος, η κυρία Αλγγελίκα Μιλινάρ, η κυρία Κάλλας την εκπροσωπεί. Ναι, ευχαριστώ. Η σκιώδηση εισηγήτρια χαιρετίζει την απόφαση του εισηγητή να υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν για ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα, είναι ένα εξαίρετο μήνυμα προς την επιστημονική μας κοινότητα και ένας καλός τρόπος να γιορτάσουμε την επέτειο της συμφωνίας αυτής στην επεξήγηση ο εισηγητής ε, ε, δίνει έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ που είναι ο μόνος μας ε, εταίρος από τις μη συνδεδεμένες χώρες ο οποίος έχει θέση στο πλαίσιο ορίζοντας 2020. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ανοιχτή τη συνεργασία ως μια γέφυρα για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις εθνικιστικές τάσεις μια τέτοια έντονη στιγμή στις σχέσεις μας. Ε, είμαστε υπέρ των προγραμμάτων ε, γιατί ενισχύεται πλήρωση η συνεργασία των δύο μερών και υπάρχει εφαρμογή προγραμμάτων σε στρατηγικούς τομείς. Επίσης υπάρχει μια έκθεση του παρατηρητηρίου των ΗΠΑ το 2016 ε, το σύστημα της καινοτομίας ε, θεωρήθηκε το πιο συνεκτικό στον κόσμο, όμως ε, κινδυνεύει από τις τάσεις στην χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί υπό την τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τα προβλήματα επίσης αυτά σε επίπεδο δημοσιονομικό ε, στην ουσία ε, βγήκαν στον τύπο πρόσφατα. Φαίνεται ότι ε, σιωπηρός η είπα, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση από την πλευρά της ΝΑΣΑ για τέτοια θέματα. Φαίνεται λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μια μεσοβραχυπρόθεσμη λύση για να μπορέσουμε να έχουμε τους πόρους που θα μας βοηθήσουμε να συνεχίσουμε την έρευνα σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς τομείς που αλλάζουν την καθημερινή μας ζωή και την επίπτωση στο περιβάλλον. Τέλειωσε ο χρόνος, με ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν πιστοί στο χρόνο. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ και την κυρία Νίμπλερ που παρακολουθεί όλες μας τις συζητήσεις και δεν μας ε, ενοχλεί στο μεταξύ με τις ιδέες της. Και τώρα τον λόγο στον κύριο Τάισεν από την Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, ευρωβουλευτές που μίλησαν σήμερα το πρωί. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό διακανονισμό. Είναι σημαντικό να συνεχίσει γιατί μας δίνει ένα πολιτικό πλαίσιο για τον διάλογο σχετικά με τους στόχους που θέλουμε να δημιουργήσουμε τους κοινού στόχους μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΥΠΑ. ΕΕ. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, θα στοχεύσουμε τη στρατηγική μας στις παγκόσμιες προκλήσεις που και οι δύο αντιμετωπίζουμε παρά τις ε, συγκεκριμένες δυσκολίες ε, που ανέφεραν οι συνάδελφοι ε, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών στη ΣΥΠΑ. Αυτό έχει θέσει τα θεμέλια για την συνεργασία μας τα επόμενα πέντε χρόνια και μας πάει στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Έτσι λοιπόν ε, είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο που συμφωνεί να επιταχύνει τη διαδικασία, να επιταχυνθεί δηλαδή η εξέταση αυτής, ε, αυτού του σχεδίου σύστασης και αδειμονώ για τον Ιούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Με χαρά μου θα δω μια σύναψη των αποτελεσμάτων υπέρ αυτής της συνεργασίας ως τώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο, θα ήταν όμως πολύ ενδιαφέρον. Χάρη στις προσπάθειές μας να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια τέτοια απλή σύνοψη για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις προσπάθειές μας. Και τώρα ο συγκητής, ο κύριος Πάξας, μπορεί να κάνει ε, κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους και, την εκπρόσωπο, και στον εκπρόσωπο της Επιτροπής που υποστηρίζουν την έκθεση και την παρουσίασή μου να δώσω έμφαση για άλλη μια φορά στο γεγονός ότι η συνεργασία σε τομείς επιστήμης και τεχνολογίας μεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντική. Καλό θα ήταν λοιπόν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή τη. Σα ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά και θεωρώ ότι αυτή η έκθεση θα είναι υποφελής για την επόμενη πενταετία. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Προθεσμία είναι 23 Μαΐου 2018 το μεσημέρι, 12 ε, η ώρα δηλαδή, για τις τροπολογίες. Όπως είπα, 12 το μεσημέρι, 23 Μαΐου, η ψηφοφορία στην Ήτρε 19 Ιουνίου και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το προχρονοδιάγραμμα που μας ζήτησε να παρακολουθήσουμε η Κομισιόν. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Γενικό Διευθυντή για το Δίκτυο Επικοινωνιών περιεχομένου και τεχνολογίας, τον κύριο Βιόλα, ο οποίος τρέχοντας μπαίνει στην αίθουσα ε, για να συζητήσει μαζί μας ε, και να μας παρουσιάσει τις εξέχουσες απόψεις του για τα θέματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη και τον, ε, το τελεία EU τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαδίκτυο. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη της Επιτροπής ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω. Είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα. Βλέπετε σήμερα στη Σόφια οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διπνήσουν και ένα από τα βασικά θέματα του δείπνου είναι η ψηφιακή καινοτομία. Θα είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση πολιτικής σχετικά με το καθεστώς της ψηφιακής ενίας αγοράς, τις σχετικές προτάσεις που βρισκόμαστε. Η παρέμβαση μου λοιπόν είναι πολύ επικαιρή σήμερα. Υπάρχει κάτι που πάντα λέω και που βέβαια εφαρμόζεται όχι μόνο, ε, δεν το λέω μόνο λόγω ευγενία, αλλά ευχαριστώ πράγματι την Ήτρε για το έργο της, για όσα κάνει αυτή η Επιτροπή για να προωθήσει την ε, ψηφιακή ενιαγορά, κυρίως αυτή την εποχή. Δεν είναι κάτι που λέω από ευγένεια ε, και γίνεται από ευγένεια, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πολύ εντατικές εργασίε της Επίτροπή Ήτρε Έχουμε σημαντικές πρόοδους στα βασικά χαρτοφυλάκια της ψηφιακής ενίας αγοράς. Συλλογικά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε δώσει μια ενία αγορά στους πολίτες. Χωρίς σύνορα, οι πολίτες μπορούν να κινούνται στην Ευρώπη χωρίς να πληρώνουν τέλη περιαγωγής, να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για να παρακολουθήσουν το περιεχόμενό τους χωρίς ε, γεωγραφικό αποκλεισμό, και στο τέλος του έτους θα μπορούν να ψωνίζουν στο διαδίκτυο τους περιορισμούς. Αυτό είναι επίτευγμα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι απλώς η αρχή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή είναι η επιφάνεια. Υπάρχουν διάφορες σημαντικές μεταρρυθμίσεις της ενιαίας αγοράς που πρέπει να ολοκληρωθούν και θα τις αναφέρω όχι αξιολογώντας τις, ε, απλώς όπως έρχονται στο μυαλό μου οι προτεραιότητες. Μεταρρύθμιση των κανόνων τηλεπικοινωνίας. Ελπίζουμε συνομοθέτης να μπορεί να καταλήξει τελική συμφωνία μέχρι τον ε, Ιούνιο, οι συνομοθέτες να βρουν λύση και αυτό θα δώσει σημαντική όθηση στην ενιαία αγορά. Η νέα πράξη για την κυβερνοασφάλεια θα δώσει στην ενίσα μόνιμη εντολή και θα υπάρξει και ένα πλαίσιο πιστοποίηση. Ελπίζουμε και αυτό να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο του έτου. να υπάρξει συμφωνία μέχρι τότε. Συνεχίζονται οι εργασίες στον τομέα των οπτικουστικό. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίε σε αυτή την Επιτροπή με συμφωνία για τη νέα οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Συνεχίζεται το έργο όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, τα πνευματικά δικαιώματα. Χρειάζεται κάποια δουλειά όσον αφορά τον κανονισμό ΚΑΠΣΑΤ ε, και την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα. Μακροσκελής ο κατάλογος, δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς σε αυτόν. Θα επικεντρωθώ σήμερα στα πεπραγμένα του Απριλίου και αρχές ε, αρχών Μαΐου. Τον Απρίλιο παρουσιάσαμε σημαντικό πακέτο με προτάσεις για την ψηφιακή ενή αγορά και αρχές Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκινώντας από το πακέτο του Μαΐου, διότι αυτά είναι αλληλένδετα όσον αφορά τα ψηφιακά θέματα. Να τονίσω ότι από τις πολλές προτάσεις μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τεχνητή νοημοσύνη και τη σχετική ανακοίνωση. Είναι ανακοίνωση περιπολιτικής. Παρουσιάζει τις ιδέες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να ακολουθήσουμε ευρωπαϊκή προσέγγιση τεχνητή νοημοσύνη που θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος, τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι επιτυχία, μια επιτυχία για την Ευρώπη. Οι εταιρείε μας, τα πανεπιστήμια μας, οι νεοφείς εταιρείε μας να ενστερνιστούν την τεχνητή νοημοσύνη και να είναι στην πρώτη γραμμή. Είμαστε στην πρώτη γραμμή στην Ευρώπη της ρομποτικής κατά παρελθόν, χάρη στο πρόγραμμα Horizon και στο προηγούμενο πλαίσιο Δυστυχώς η επιχειρηματικότητα της Ευρώπης τώρα κινείται πιο αργά από τις άλλα του κόσμου. Και κάποια από τα κοσμήματά μας όσον αφορά τη ρομποτική έχουν αγοραστεί από μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα ανακαλύπτονται στην Ευρώπη και θα παραμένουν στην Ευρώπη διότι πιστεύουμε ότι τεχνική, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι καλό. Βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των πολιτών, στην ιατρική, στις δημόσιες υπηρεσίες, στην παραγωγή. Ο τόπος εργασίας γίνεται ασφαλέστερος και δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες. Βέβαια, και αυτό ανοίξει το δεύτερο πυλώνα, υπάρχουν και προβλήματα. Η τεχνική η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει εις τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμεθα και θα εργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίζουμε κάποια κοινωνικά προβλήματα και αυτό χρειάζεται προσεκτική εξέταση όσον αφορά τις εξέτασεις του εργατικού δυναμικού, τον κίνδυνο για το εργατικό δυναμικό, αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Σημαντικό το το. Εργόδιο τεχνητή λοημοσύνη θα μεταμορφώσει πάρα πολλούς τομείς. Τρίτος πυλώνας της στατικικής. Διοντολογικά θέματα και νομικά ζητήματα σχετικά με τη τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρώπη μπορεί να είναι μοναδική όσον αφορά την προάσπιση των αξιών της και των κεκτημένων της. Να εξασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισάγεται στην κοινωνία μας με ένα βιώσιμο τρόπο, με ένα διαφανή τρόπο, ε, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν θέλουμε τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα αποφασίζουν για το μέλλον των ανθρώπων. Δεν θέλουμε ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνης που θα ελέγχει τους ανθρώπους που θέλουν, έχουν, ε, να πάρουν, θέλουν να πάρουν κάποιο δάνειο, να βρουν κάποια θέση εργασία ή να μπουν σε πανεπιστήμιο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο στην κοινωνία μας. Το βλέπουμε ότι εκφράζονται κάποιες ανησυχίες. Βλέπουμε ότι κάποια συστήματα που έχουν εισαχθεί στην Κίνα τι κάνουν για τα δάνεια, χορήγηση δανείων, πώς γίνεται η δίθυση των υποψηφίων εδάνειων όσον αφορά τα μικροδάνεια που πηγαίνουν στι οικογένειε, ε, Όπως σας είπα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πολύ επωφελής και να βελτιώσει την ποιότητα ζωή των πολιτών, ταυτόχρονα όμω, πρέπει να αναπτυχθεί με έναν τρόπο που σέβεται τις αξίες μας και την ένωμη τάξη μα και τι ε, ηθικές αξίε. Αν καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, είναι πεπισμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρώπη μπορεί να βρει μοναδική θέση και να ακολουθήσει το δρόμο της για τη βιώσιμη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουμε το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σαν μια λογική συνέχεια της ανακοινώσεως για την τεχνητή νοημοσύνη στις 2 Μαΐου ανακοινώσαμε το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, σαν τμήμα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη ανήκει σε ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο που αφορά την ενιαία αγορά, ε, την ψηφιακή ενιαία αγορά και την καινοτομία. 180 δις ευρώ αφορά αυτό που θα διτεθούν για την ε, ριζική αλλαγή που θα είναι υποφελής για την κοινωνία. Εντός του κεφαλαίου αυτού θα έχουμε το νέο πρόγραμμα πλαίσιο ορίζον Ευρώπη και το νέο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη και η συνέχεια του ΣΕΦ. Ο τρόπος που διοργανώνουν τα πράγματα είναι το ΣΕΦ. Θα ασχολείται με θέματα υποδομών. Θα θυμόσαστε ότι το ΣΕΦ είναι κάτι ανάμεικτο. Υποδομές και υπηρεσίες. Θα συνεχιστούν όλες οι δραστηριότητε του ΣΕΦ στα πλαίσια του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και το πρόγραμμα της Ψηφιακή Ευρώπη θα επικεντρώνεται επί τη δυνατότητα που έχει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τα τρία βασικά προβλήματα που αφορούν τον ψηφιακό τομέα. Τη δυνατότητα να έχουμε πολύ μεγάλου υπολογιστέ, πολύ δυνατού υπολογιστέ, υπερ, και να έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη με δημόσιε υπηρεσίε που έτσι θα αποφεληθούμε από τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια. Στα θέματα κυβερνοασφαλείας θα δούμε και μια πρόταση για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αριστείας όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια για να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data, ε, νέα τεχνολογία για να έχουμε ασφαλέστερο οικοσύστημα, πιο ανθεκτικό. Αυτά εν κατακλείδη είναι αυτά που θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως μερικά λόγια να πω για το υπόλοιπο πακέτο. Κάτι πολύ συναφές, θέλουμε να δημιουργήσουμε ενιαίο χώρο δεδομένων στην Ευρώπη έναν ενιαίο χώρο όπου οι ίδιοι κανόνες περιδιωτικότητας θα ισχύουν, οι ροές των δεδομένων θα την χάνουν εγγυήσεων και ταυτόχρονα θα μπορούν να διατηρούνται αυτά τα δεδομένα. Τεχνητή νοημοσύνη επί έτη υπάρχει από πολύ παλιά. Ήμουνα φοιτητή όταν ξεκίνησε και δοκιμάστηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που κάνει τεχνητή νοημοσύνη κάτι επαναστατικό είναι η πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Τα δεδομένα θα πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη, να συλλέγονται εκεί και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα με σωστό τρόπο για τα πάντα. Τα περισσότερα δεδομένα σήμερα αποθηκεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό βέβαια βάζει την Ευρώπη ε, σε πολύ μειονεκτική θέση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό προτείναμε ένα πακέτο για τα δεδομένα που εξετάζει την αδιάθρωση οδηγία του PSI, μία από τις επιτυχίες της Επιτροπής σας και της Ευρώπης είναι η ανοιχτή πολιτική για τα δεδομένα στην Ευρώπη, για ανοιχτά στοιχεία. Τώρα θέλουμε να παγιώσουμε αυτή την πολιτική για τα ανοιχτά δεδομένα, να δούμε τι γίνεται με τις κοινοφελείς υπηρεσίες, να δούμε με ποιο τρόπο η διοίκηση ασχολείται με τα open data. Διότι όσο περισσότερα ελεύθερα ανοιχτά στοιχεία έχουμε, τόσο περισσότερο θα μπορούν οι επιχειρήσεις να τα χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη Στείλαμε ένα σαφές μήνυμα, δεν θέλουμε να ρυθμίσουμε την ανταλλαγή των στοιχείων μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δώσαμε κάποιους προσανατολισμούς, ήπιους προσανατολισμούς σχετικά με τους καλύτερους τρόπους ε, αντιμετωπίσεως του θέματος. Αυτό βέβαια φαντάζομαι θα αποτελέσει και ένα τμήμα των συζητήσεων. Επίσης ε, προτείναμε κανόνες ε, δικαιοσύνης, δικαίου όσον αφορά τις πλατφόρμες, ώστε οι πλατφόρμες όσον αφορά τις Ευρωπαϊκής επιχειρήσης, εφαρμόζουν κανόνες διαφανείας που απαιτούνται για θεμητές επιχειρηματικές σχέσεις και μηχανισμοί αποζημίωσης ε, είναι αποτελεσματικοί αν κάτι πάει λάθος και θα, θα ρυθμίσει το θέμα της Ευρώπης με ο κατάλογος Πρόεδρε. Ίσως τα μέλη σας να έχουν ερωτήσεις για άλλα στοιχεία του πακέτου για να μην χρονοτριβώ λοιπόν θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο κατά ένα λεπτό περάσατε το δεκάλεπτο για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Βέβαια, έχουμε 8 χαρτοφυλάκια στο πακέτο. Ε, βλέπουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινό χώρο δεδομένων στην Ευρώπη, ε, οδηγία για τη χρήση των δεδομένων, για τις πληροφορίες του δημόσιο τομέα, για πρόσβαση και διατήρηση επιστημονικών πληροφοριών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κανόνες για την διαβίβαση στοιχείων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ευρύτατο πεδίο εφαρμογή, ε, πολλαπλά στοιχεία και υλικό ε, που αναλύεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Και δύσκολο να συνοψιστούν όλα αυτά σε ένα δεκάλεπτο. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε οι συντονιστές οι αντικαταστάτες τους. Ο καθένας έχει ένα τρίλεπτο στη διάθεσή του. Άλλα ενδιαφερόμενα μέλη μετά θα έχουν ένα λεπτό ο καθένας. Δεν είμαστε και πολλοί παρόντες, οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, διότι ο καθένας μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. ΕΛΚ. Η κυρία Καστίγιο Βέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ στα τρία λεπτά που έχω χρόνο και νομίζω ότι μπορεί να τα πω και πιο γρήγορα γιατί ο χρόνος πιέζει. Είναι προφανές πως δεν είναι καινούριο το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι ότι υπάρχει εδώ και πάντοτε, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μια έννοια την οποία συζητάμε. Και αν δείτε μόνο τον αριθμό των ταινιών που έχουμε παρακολουθήσει, που τις τελευταίες δεκαετίες Ε, βασίζουν την υπόθεσή τους σε τεχνητή νοημοσύνη με τα πιο εξελιγμένα των τελευταίων ετών είναι ξεκάθαρο που βρίσκεται το θέμα. Όπως είπατε κι εσείς, το θέμα των ψηφιακών δεδομένων έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, οι τεχνολογίες ψηφιακές έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που οι επιπτώσεις στην κοινωνία είναι τεράστιες και τελείως διαφορετικές από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωση αυτή για τις μελλοντικέ εξελίξεις στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής. Καταρχήν, μια γενικότερη ε, ερώτηση που έχει να κάνει με το πολιετές πλαίσιο χρηματοδότησης και τις συζητήσεις για το επόμενο πλαίσιο, ε, πρόγραμμα πλαίσιο στην έρευνα. Για την τεχνητή νοημοσύνη, τι προβλέπετε εκεί. Αναφερθήκατε σε διάφορα στοιχεία, αλλά θα ήθελα αν μπορείτε να μου δώσετε λεπτομέρειες. Δεύτερον, η ανακοίνωση μιλά για προτάσεις οι οποίες ε, θα γίνουν στα πλαίσια του επόμενου πολίτης πλησίου θα δώσουν ενισχυμένη στήριξη για την απόκτηση ε, εξελιγμένων ε, τεχνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα δεξιοτήτων στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς θα γίνει αυτό, τι έχετε προβλέψει. Μετά. Τρίτο. Τι είναι αυτά τα regulatory sound boxes που αναφέρεται στην ανακοίνωση που θα στηρίζουν στις μεταφορές, στην βιομηχανία, στον κλάδο υγείας, στα ε, γεωργικά και στα τρόφιμα, αυτά τα IT ε, hubs. Και πιο συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη και το ψηφιακό πακέτο τι μέλλον θα έχουν. Θα καταθέσετε περισσότερη νομοθεσία ήδη σε αυτή τη θητεία ή απλώς μέσω αυτών προσπαθείτε να βρείτε ένα διάδρομο προσγείωσης για την επόμενη θητεία. Λόγω και των χρονικών πιέσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, γιατί δεν έχει μείνει ούτε κανένας χρόνος μέχρι τις εκλογές. Έχετε κάτι να πείτε? Η ομάδα μου πολύ θα ήθελε να το ακούσει. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος είναι να συνοψίσουμε ε, όλες τις ερωτήσεις μαζί, δηλαδή να τις ε, συλλέξουμε όλες τις ερωτήσεις και να απαντήσετε ε, συνοπτικά σε όλους. Ο κύριος Ζωρίνιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον, καλωσορίσω τον Γενικό Διευθυντή και να τον συγχαρώ για το πόσο φιλόδοξο είναι το πρόγραμμα αυτό. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να απαντήσετε σε μία ερώτηση. Χτες έληξε η πληθυσμία για την προεγραφή των Δήμων στην ε, πρωτοβουλία Wi-Fi for You. Και ήταν μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. δική μου χώρα το 75% των Δήμων προσπάθησαν να κάνουν αυτή την προεγγραφή. Και αυτό αποδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό. Η κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη είναι έτοιμη για να ξεκινήσει τη μάχη για τη νέα ψηφιακή επανάσταση. Όμως, ταυτόχρονα, η καθυστέρηση στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος που θα ήταν ο πυρήνας αυτών των προσπαθειών αποδεικνύει ότι η Ευρώπη χρειάζεται να προετοιμαστεί καλύτερα και πιστεύω πως ε, μία από τις καλύτερες πολιτικές που θα μπορούσαμε να φανταστούμε είναι ακριβώς αυτή. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να χάσουμε την αξιοπιστία μας στη στιγμή της εφαρμογής. Οι ιδέες μας είναι πάντα εξαιρετικές, αλλά θα πρέπει να τις εφαρμόζουμε κιόλα με τον ίδιο εξαιρετικό τρόπο. Πρέπει να δώσουμε σταθμισμένες και βιώσιμες απαντήσεις, οι οποίες θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή. Και οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τι επιθυμίε των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν για να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα που θα μα επιτρέψει να πρωταγωνιστήσουμε σε μια ε, κοινωνία ε, ανθρώπων και μηχανών, να γίνει μια πιο αξιοπρεπής κοινωνία, μια κοινωνία ανοιχτή και όχι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ανθρώπου και μηχανών ε, άνηση που δεν θα προσφέρει ευκαιρίες. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνετε. Σας καλωσορίζω μια φορά ακόμα. Είναι μια νέα ευκαιρία με την αύξηση ε, του προϋπολογισμού ε, για την ψηφιακή καινοτομία αυτά τα επιπλέον ένα δις και θα πρέπει με 100 εκατομμύρια και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να βρει μια ταχύτητα πλεύσης η οποία ε, θα μας επιτρέψει να μεταμορφώσουμε την ψηφιακή πραγματικότητα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Άλλος, από τους Σκιώδης, ποιος θέλει να πάρει το λόγο για να το σχολιάσει. Οκ, η κυρία Νίμπλερ, η οποία σίγουρα έχει προετοιμάσει τα σχολεία της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πάντα έχω αξιόλογα σχόλια, θα ήθελα και εσείς να το συμμερίζεστε. Ε, θα πω ότι μας έχετε δώσει μια γενική επισκόπηση σχετικά με τα όσα ε, ε βάσει της δράσης της γενικής σας διεύθυνσης στο τομέα της ψηφιακής αγοράς. Νομίζω ότι στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε καλό δρόμο σχετικά με κάποιες προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης και με το αντίστοιχο πλαίσιο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ε, συναδέλφους να ε, περάσουν τα διάφορα εντοσχέτους τους και να τα κλείσουν ε, μέσα σε αυτή την νομοθετική περίοδο. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες ερωτήσεις για την, ε, για την νοημοσύνη, την ανακοίνωση, την έχω δει στα πεταχτά. Ε, νομίζω ότι σε αυτή την ανακοίνωση υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, ποιο είναι το κλειδί έτσι ώστε εμείς στην Ευρώπη να παίξουμε σημαντικό ρόλο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, κι άλλο ένα ερώτημα για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί υπάρχει τεράστια συζήτηση στη χώρα μου για αυτό το θέμα. Πόσο θα επιτρέψουμε ε, εταιρείε όπως η Google, επιχειρήσεις που ξέρουν, που έχουν την τεχνολογία κλειδί, την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία, να εξαγοράζονται από τρίτες χώρες. Ε, έχει να κάνει με τις εμπορικές ε, συμφωνίες, όμως πώς θα προστατεύσουμε εμείς την βιομηχανία μας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε, να υπάρχει ένα ελάχιστο στάνταρ εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα πρέπει να τηρούν και οι τρίτες χώρες. Άλλο ένα ερώτημα για τις ε, δημιουργικές βιομηχανίες, creative industries. Είναι μεγάλη η βιομηχανία αυτή και σε εμάς. Ε, προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών. Ε, θα θέλαμε κάποιες προτάσεις σύντομα να μας παρουσιάσετε γι' αυτό και τέλος για τις ψηφιακές δεξιότητες, digital skills. Στην Ευρώπη έχουμε την ανάγκη να φτάσουμε στο αντίστοιχο επίπεδο ακόμα. Οι γυναίκες ιδιαίτερα δεν έχουν όλες αυτές τις δεξιότητες. Ε, θα πρέπει να, κάνουμε, λοιπόν, να έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες συγκεκριμένα θα προσπαθήσουν να κινητοποιήσουν τις γυναίκες και θα δώσουν τα κίνητρα στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν αυτό το δυναμικό ειδικά των γυναικών ας πούμε με την δημιουργία νεοσύστατων επιχειρήσεων, startups ε, ή ε, με τεχνικά επαγγέλματα. Ε, σε αυτούς τους τομείς βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ενίσχυση για να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το δυναμικό. Τώρα για τον κανονισμό σχετικά με τις πλατφόρμες υπάρχει μια τεράστια συζήτηση. Νομίζω ότι η πρότασή σας δεν είναι και τόσο φιλόδοξη. Θα θέλαμε να είναι πιο φιλόδοξη. Ε, και να μην είναι τόσο light regulation. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις ε, ετέθησαν και ο, ο Γενικός Διευθυντής φαντάζομαι ότι θα μας δώσει και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Ποιος άλλος θέλει να μιλήσει, η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πολλή δουλειά. Και ο δικός σας κλάδος στις νέες ε, πολυετής προοπτικές νομίζω ότι τα πάει θαυμάσια και σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι γιατί πια έχουμε την οριμότητα για την ψηφιοποίηση να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Εγώ συνήθως δεν είμαι τόσο ενθουσιώδης αλλά Θέλω να συνδυάσω αυτή την ε, παρατηρήση που κάνω με την παρότρινση να βρούμε κάποιες λύσεις. Λύσεις τις οποίες ε, να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Κλίμα, ενέργεια, να δούμε πώς εκεί θα βάλουμε και την ψηφιοποίηση. Και επίσης την ηλεκτρονική υγεία ή health γιατί για το μέλλον. Να σας πω πως δεν είναι πολύ μεγάλο το, το πρόγραμμα υγείας που προτείνεται και αν το συνδυάσουμε με το θέμα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες υγείας ε, και την σχετική ανακοίνωση, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα συνεργαστούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί. Εγώ δεν είμαι γιατρός, είμαι μηχανικός και ανησυχώ αν όλες αυτές οι πληροφορίες Ε, συλλεχθούν όχι από ε, το δημόσιο αλλά από ιδιωτικές επιχειρήσεις τι προστασία ε, θα έχουν αυτά τα δεδομένα. Και τι θα γίνει η φαρμακοβιομηχανία για ανθρώπους που έχουν ψυχικά προβλήματα για παράδειγμα θα συνταγογραφεί υπερβολικά. Βλέπουμε τι γίνεται με τα οποία τι για παράδειγμα. Γιατί πολλές φορές οι ανάγκες χρησιμοποιούνται μέσω του κατάλληλου μάρκετινγκ. Οπότε η ιδέα μου είναι η εξή. Τα δεδομένα για την υγεία θα είναι πλέον ε, δημόσια, θα τα μοιράζονται οι δήμοι, τα νοσοκομεία, το κράτος, αλλά και οι επιχειρήσει του κλάδου. Γιατί υπάρχει και το θέμα ε, της ε, ιδιωτικής ζωής. Και το είπε και ο Μακρόν όταν πήγε στην Γερουσία ε, στην Ουάσιγκτον. Θα πρέπει παρόλα αυτά να βάλουμε κάποιους ε, κανόνες όσο και αν δεν θέλουμε να κάνουμε ε, να μην κάνουμε υπερβολικές νομοθετικές προσπάθειες. Οπότε τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει κάποιο είδους εγκάρσιο τρόπο σκέψης για τα προγράμματα αυτά και για την πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται να ρυθμίσουμε κάπως Θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε να χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες και θέλω να χρησιμοποιούνται και από το δημόσιο. Θα έπρεπε κάθε πόλη να χρησιμοποιεί τέτοιες πλατφόρμες, αλλά ο ανταγωνισμός τι σημαίνει. Ότι παρέχουμε πληροφορίες στους ε, επιχειρηματίες ή ότι θα περνάει κάποιο είδου έλεγχο και ότι θα έχουμε την πληθώρα ε, προϊόντων στην αγορά που είναι αυτέ που χρειαζόμαστε. Οπότε χρειάζεται να σκεφτούμε πάρα πολύ και τα θέματα τα ηθικά ε, και εμείς ως Ευρωπαίοι και ως ε, Ευρωβουλευτές θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Τόσες πολλές και τόσες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Να προσθέσω και εγώ τη δική μου. και να σας πω πως κάτι το οποίο είναι σημαντικό για κάθε πολίτικη, για κάθε πολίτη, είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στο, στην για παράδειγμα, είναι τεράστιο πρόβλημα με τα μικρά χωριά, όπου πολλές φορές δεν έχουν καν τη διάθεση να έχουν ίντερνετ. Με αυτά τα πολύ μικρά χωριά. Και ίσως αυτό είναι και το πρόβλημά μας. ασφάλεια δεδομένων αφενός και ανοιχτά δεδομένα από την άλλη, open data. Σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων όλα αυτά Ξέρετε ότι πάρα πολλά δεδομένα αποθηκεύονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνουμε για να τα προστατεύσουμε και για τον κυβερνοχώρο και για να μην εξαρτώμεθα από εξωτερικούς παράγοντες. Επίσης, τυποποίηση, προστασία της βιομηχανίας, της δικής μας βιομηχανίας. Για παράδειγμα, στη Χαλιβουργία χρησιμοποιούν πάρα πολλά δεδομένα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εξυπηρέτηση ε, πελατών, έχουν να κάνουν και με την ίδια τη γραμμή παραγωγής. Για παράδειγμα, ε, θερμοκρασίες, ε, ατμοσφαιρική πίεση, όλα αυτά θα πρέπει να σχετιστούν κάπως με την ε, προστασία που θα προσφέρουμε. Και εμείς όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να συλλέξουμε τεράστιο αριθμό ε, δεδομένων, να τα αξιολογήσουμε. Μπορούμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα καταρχήν να τα μοιραστούμε και δεύτερον να τα προστατεύσουμε. Πολλές φορές δεν μπορείς καν να επισκεφτείς την Υψικάμινο γιατί δεν έχεις την πραγματογνωμοσύνη. Και παρόλα αυτά ξέρεις πως πρέπει να πας γιατί εκεί υπάρχει κάτι καινούριο. Οπότε ποια είναι η γραμμή που χωρίζει την προστασία και ε, τα ανοιχτά δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πόσα λεπτά έχω για να απαντήσω. 20 λεπτά. Α, πολύ ωραία. Άρχισα να ε, αισθάνομαι ότι θα ήταν τροπή να απαντήσω συνοπτικά σε τόσο βαθιές ερωτήσεις. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ερωτήσεις. Μπήκανε σε βάθος και θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις ε, όσο καλύτερα μπορώ. Θα ξεκινήσω με τη σειρά, με την κυρία Ντελ το πρώτο θέμα που θέλω να ξεκαθαρίσω έχει να κάνει λίγο με το χρονοδιάγραμμα ε, το πακέτο του Απριλίου και της άσκησης του πι Τον Απρίλιο έχουμε το πακέτο, μετά η Κομισιόν θα σας δώσει όλη την εικόνα για το πι και αρχές Ιουνίου θα έχουμε την πρόταση προγραμμάτων που έχει οθετήσει το Κολέγιο των ε, Επιτρόπων. Οι σχετικές προτάσεις για τον ψηφιακό τομέα θα είναι ε, το νέο πρόγραμμα Νέος Ορίζοντας, ε, το, η ψηφιακή Ευρώπη, συνδέοντας την Ευρώπη και η νέα ε, δημιουργική Ευρώπη, New Creative Europe. Αυτές είναι οι βασικές επενδύσεις στις οποίες θα επικεντρωθούν οι προτάσεις. Το πρόγραμμα Digital Europe θα έχει μία δίδυμη πρόταση σε επίπεδο εκτέλεσης. Θα είναι αυτός ο κανονισμός ο οποίος δημιουργεί το ε, δίκτυο των κέντρων ε, ικανότητα στον κυβερνοχώρο, Cyber Competence Center. Αυτό θα εγκριθεί αρχές Ιουνίου από την Κομισιόν, από ό,τι φαίνεται, σε δύο συνεδριάσεις αρχές Ιουνίου και φυσικά θα είμαι πανέτοιμος να επανέλθω μόλις ε, κατατεθούν οι προτάσεις και να σας απαντήσω λεπτομερώς σε οτιδήποτε θέλετε να ξεκαθαρίσουμε στην Επιτροπή σας. Αυτά γενικά. Τώρα, κάποια πράγματα μπορώ να τα προβλέψω, γιατί υπήρξε η ανακοίνωση της Δευτέρας Μαΐου για το δέλτα. Η τεχνητή νοημοσύνη. Πού θα βρίσκεται, αυτό ρώτησε η κυρία Ντεκαστηγιό, όσον αφορά τους βασικούς πόρους θα είναι στο νέο πρόγραμμα Ορίζοντας, New Horizon. Ε, τώρα σε επίπεδο εφαρμογών, δημιουργία ικανοτήτων, δημοσίων υπηρεσιών, δεξιοτήτων θα είναι στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη και σε επίπεδο καλύτερης προστασίας ε, των παγίων μας ε, θα είναι ε, στα κέντρα για την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Εκεί θα δούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα έχει βασικά πέντε κλάδους. Big Data και Super Computing, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συνέχιση των σημερινών ασφαλών δραστηριοτήτων σε επίπεδο ψηφιακών δραστηριοτήτων και τις προχωρημένες δεξιότητες. Δεξιότητες ε, τώρα. Τι είναι. Έχουμε ευθύνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να ενισχύσουμε τη συζήτηση για τις δεξιότητες ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα κράτη-μέλη, αλλά και να κάνουμε πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο θεωρούμε ότι οι προχωρημένες ψηφιακές ε, δεξιότητες που σχετίζονται με το big data, την τεχνητή νοημοσύνη, τα super computers ε, είναι σε σπάνιδα στην Ευρώπη, είναι μεγάλο πρόβλημα και χρειαζόμαστε τα πανεπιστήμια και τα κέντρα γνώσης να συνεργαστούν. Όσο πιο κάτω πάμε σε επίπεδο δεξιοτήτων που πρέπει να εφαρμοστούν στο σύστημα παραγωγής υπηρεσιών, παντού δηλαδή η βασική γνώση των ψηφιακών δεξιοτήτων όσο πιο κάτω πάμε τόσο πιο μεγαλύτερη ευθύνη έχουν τα κρατημέλη, οι περιφέρειες, οι τοπικοί θεσμοί και είναι λιγότερο ευθύνη κεντρικών προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν ε, σε αυτό επικεντρώνεται ε, το ε, πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη στις προχωρημένες δεξιότητες αλλά γενικά η συζήτηση για τις δεξιότητες, τις βασικές δεξιότητες είναι μια συζήτηση που συνεσχίζεται αλλά δεν πρέπει να το παρακάνουμε ε, σε πράγματα που τόσο ή γίνονται καλύτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εμείς μιλάμε για τις προχωρημένες δεξιότητες τα regulatory sound boxes. Είχαμε μία ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της οικονομίας, το λεγότερο FinTech. Ε, αυτά τα εργαλεία είναι σχετικά παρόμοια. Ε, συνοπτικά υπάρχει ένας τοπικός ρυθμιστής που για λίγο χρονικό διάστημα, λίγους μήνες, ένα χρόνο, θέτει κάποιες νομικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή νέων οικονομικών υπηρεσιών. Ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη, ο τοπικός ρυθμιστής, η ρυθμιστική αρχή θέτει κάποιες απαιτήσεις που δεν είναι και τόσο ουσιαστικές, αλλά βελτιώνουν την καινοτομία. Γι' αυτό είναι και προσωρινές και δίνονται κυρίως στη startup και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Φυσικά, αυτή η ιδέα μπορεί να αναπαραχθεί σε πολλούς άλλους τομείς. Κατά περίπτωση, λοιπόν, η ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίσει πώς θα διευκολύνει την καινοτομία. Η τελευταία ερώτηση ήταν εάν χρειάζεται να έχουμε περισσότερη νομοθεσία μετά τις προτάσεις του δελτα την ψηφιακή Ευρώπη και τα competence centers δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές άλλες ψηφιακές, ε, συγγνώμη, νομοθετικές προτάσεις για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Γιατί λογικά θα έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο και θα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που θα πρέπει να γίνουν για να διασφαλίσουμε ότι θα μπει σε εφαρμογή αυτό που έχουμε θεσπίσει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα έχουμε κάποιες βασικές νομοθετικές πράξεις εκτός αν υπάρχει κάποια εκτακτή ανάγκη. Ο κύριος Τζορίνιο μίλησε για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για μας, Wi-Fi for Europe. Εχθές γιόρτασε την πρώτη μέρα διανομής των voucher. Από την ημέρα που ξεκίνησε είναι πολύ επιτυχημένο το πρόγραμμα. Και δεν πίστευαν όλοι στην επιτυχία, το θυμάστε κύριε Ζουρίνιο. Στο Συμβούλιο, ειδικά κάποια κράτη-μέλη, πραγματικά θεωρούσαν ότι δεν, δεν θα ενδιαφέρονταν οι δήμοι. Όμως ε, τα νούμερα λένε πολλά. Βλέπουμε ποιοι είναι οι δήμοι που έχουν εγγραφεί και έχουν κάνει αίτηση. Και τελικά έχουμε τόσες πολλές αιτήσει που δεν έχουμε καν τα αντίστοιχα κονδύλια. Θα ανοίξουμε το θέμα λοιπόν στο δελτα. Στο επόμενο δελτα έχουμε τρία δις ε, για το προμπαντ Ευρυζωνικά. Ε, θα δώσουμε λοιπόν ε, voucher και σε άλλες μικρές οντότητες και για νέες τεχνολογίες 5G κτλ. Ναι, καθυστερήσεις υπήρξαν ίσως υποεκτιμήσαμε λίγο, υπερεκτιμήσαμε συγγνώμη, το ε, σύστημά μας για τη διανομή των micro-vouchers. Τώρα τα καταφέραμε, έχει γίνει, αλλά είναι πιο πολύπλοκο το σύστημα από ό,τι περιμέναμε. Το καλό βέβαια είναι ότι τώρα μπαίνουμε στην επιχειρησιακή φάση υπάρχουν περισσότερες παρεμβάσεις και ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται από ό,τι περιμέναμε. Πολλά ακόμα πρέπει να λυθούν. Όταν αρχίσει να τρέχει όμως το σύστημα, η επιτυχία θα φανεί σε πολλά επίπεδα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μάθημα και για το μέλλον. Αυτά που, πρέπει να θα προτείνουμε θα πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμα, ειδικά σε ψηφιακό επίπεδο. Και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό με σωστό τρόπο είναι να έχουμε καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη από την πρώτη ημέρα. Αυτό κάνουμε και με το πρόγραμμα Supercomputing. Θα το συνδέσω λίγο και με την ερώτηση της κυρίας Νίμπλερ εδώ η ψηφιακή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεράστια πρόκληση. Αν δείτε πόσο δημόσιο χρήμα διοχετεύει η Κίνα σε δραστηριότητες αμυντικές, κυβερνητικές, πραγματικά τρομάζεις. Οι ΙΠΑ συνήθως έχουν μεγάλα προγράμματα αμυντικά επίσης. Εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε τίποτα από τα δύο. Την Δευτέρα Είχα πάει στο Βερολίνο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και επέμεινα ότι υπάρχουν προκλήσεις σε επίπεδο Ευρώπης, σε αυτό το μέγεθος, όχι μόνο ε, στο μέγεθος των μεγαλύτερων κρατών μελών. Η Ευρώπη είναι όλοι μας. Είμαστε εμείς στην Ευρώπη, τα κράτη-μέλη και όλοι μας πρέπει να συνεργαστούμε. Αν θεωρούμε λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρόκληση, το επόμενο βήμα είναι να συνεργαστούμε. Είναι καλό που υπάρχουν πρωτοβουλίες από τη Γαλλία και τη Γερμανία για την ε, τεχνητή νοημοσύνη και από πολλά κράτη ε, μέλη. Γι' αυτό ζητήσαμε τον Απρίλη από τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν, να ενταχθούν σε ένα κοινό δίκτυο έτσι ώστε να ε, κάνουμε τη διαφορά. Όταν παρουσιαστεί σε τρεις εβδομάδες το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη θα δείτε ότι φυσικά προσπαθούμε να δούμε και τα βασικά αλλά και τα επιχειρησιακά ζητήματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα ε, δεδομένα ε, τα επεξεργαζόμαστε, τα χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη, ότι μένουν στην Ευρώπη και απαντώ στην ερώτησή σας Πρόεδρε. Ε, άρα θέλουμε μια έρευνα η οποία δεν είναι μόνο bottom-up δεν αρκεί η Ευρώπη μέσα από το Digital Europe θα πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση εντάξει κάναμε την έρευνα τώρα τι. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι τα super computers, είναι καινοτόμα αλλά ε, αυτή τη στιγμή ε, ε, δεν έχουμε ευρωπαϊκά super computers ε, που είναι σημαντικά για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί, γιατί δεν παρακολουθούσαμε ποτέ τις εξελίξεις όπως κάναμε με την Airbus. Εντάξει, εκεί είπαμε ότι ε, πρέπει να κάνουμε την Airbus στο Γαλιλαίο. τώρα θα γεμίσουμε και αυτό το κενό και ξέρω ότι θα έχετε μια γνωμοδότηση σύντομα για αυτό το θέμα. Οπότε η ψηφιακή Ευρώπη θα συνεχίσει, θα πάμε στην επόμενη γενεά των super computers, θα επιμείνουμε στα competence data centers για την τεχνητή νοημοσύνη ε, και εφαρμογές καινοτομίας έτσι ώστε η ε, ε, Ευρώπη να γίνει πραγματικά ψηφιακή και ειδικά να έχουμε και προχωρημένες δεξιότητες. Επίσης αναφερθήκατε σε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, δεν θέλουμε απλώς να ξεκινούν ως ευρωπαϊκές αλλά να παραμένουν ευρωπαϊκές ειδικά όταν έχουμε εξαγορές όπου η πηγή του χρήματος είναι ξεκάθαρο πως ε, ε, είναι ιδιωτικό χρήμα. Έχουμε παρουσιάσει ένα εργαλείο, το Trade Defense Instrument, ένας μηχανισμός άμυνας, εμπορικής άμυνας. Ε, έχουμε κάνει μια διαγνωστική ας πούμε μελέτη για να δούμε ε, να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια που έρχονται εκτός Ευρώπης θα μπουν κάτω από την ομπρέλα αυτού του μηχανισμού. Όταν εγκριθεί αυτό από τους επιτρόπους θα έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαγνωστικό ας πούμε στην Ευρώπη έτσι ώστε να εξετάζονται όλες οι επιχειρήσεις που θα ε, δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής ε, νοημοσύνης ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, η creative industries, η δημιουργική βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική σε επίπεδο παραγωγής ΑΕΠ. Κάνουμε αρκετά. Ό,τι και να κάνουμε, μάλλον ποτέ δεν θα αρκεί. Αν δείτε και τη μαζική χρήση των έργων, των πλατφόρμων για έργα των δημιουργών εντός και εκτός Ευρώπης, θα καταλάβετε ότι τίποτα δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει οπωσδήποτε μετά να ολοκληρώσουμε την εργασία για την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα, με όποιο τρόπο αποφασίσουν δημοκρατικά τα θεσμικά όργανα. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Ε, έχουμε τώρα όμως ε, μια δημοκρατική διαδικασία η οποία είναι και σημείο αναφορά στην Ευρώπη. Όσο δύσκολο και είναι αυτό το ζήτημα λοιπόν και η συζήτηση, γιατί είναι, θα πρέπει να φτάσουμε σε μια απόφαση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Τώρα για ό,τι θα κάνουμε στις πολιετήσεις προοπτικές θα πρέπει να δείτε ότι έχουμε προτείνει μια σημαντική αύξηση ε, των ε, ε, προγραμμάτων στα πλαίσια του Creative Europe γιατί ήταν πολύ πετυχημένο και πολλές από τις πολύ δημοφιλείς ταινίες που πήραν και ο Όσκαρ και αναγνωρίστηκαν και στις Κάνης και στη Βενετία και στο Φεστιβάλ του Βερολίνου έχουν ε, χρηματοδοτηθεί από αυτό το πρόγραμμα Media, οπότε είναι πετυχημένο. Ψηφιακές δεξιότητες. Όπως είπα, αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Ξεκινήσαμε όπως και με το Wi-Fi for You για να δοκιμάσουμε ε, το πώς έχει κατάσταση είναι κάτι το οποίο είναι δημοφιλές και μπορεί να δώσουμε υπερβολικές υποσχέσεις. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε τα, όσα θα υποσχεθούμε να τα παραδώσουμε. Και να σας πω ότι σε επίπεδο επιτρόπου εμβληματική πολιτική θεωρείται να αποκαταστήσουμε και στον ψηφιακό κόσμο την ε, ισορροπία αριθμών μεταξύ ε, φύλων και στη διαχείριση και, στα, και στις δεξιότητες, γιατί εκεί τα ποσοστά μας ε, σε γυναίκες είναι απαράδεκτα χαμηλά. Έχουμε την συνάδελφο Λορέντζα Μπουαλόντσο εδώ, που είναι ε, αρμόδια στην DigiConnect για το θέμα αυτό και εμεί οργανώνουμε μια μεγάλη διάσκεψη, μια εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, στις 19 Ιουνίου εδώ στις Βρυξέλλες για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, δηλαδή τις γυναίκες στον ψηφιακό κόσμο και θέλουμε να γίνει μια πραγματική συζήτηση με όλους και να είμαστε σίγουροι πως καταλαβαίνουμε τι πρέπει να γίνει. Αυτά τα λέω γιατί ίσως αυτός είναι ο κατάλληλος τόπος για να εμβαθύνουμε στην άποψή σας. Ρύθμιση για τις πλατφόρμες. Δύσκολα και εδώ να πετύχουμε την ισορροπία μεταξύ της επίλυσης προβλημάτων και ανησυχιών. Εμείς προσπαθούμε να καταθέσουμε ένα μέσο το οποίο θα λύνει τα προβλήματα. Δηλαδή βρίσκουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να πετύχουμε λύσεις. Επιπλέον αυτού όμως Έχουμε και τις ανησυχίες των εταιριών και των ε, μικρομεσαίων εταιριών όταν έχουν απέναντί τους μεγάλες πλατφόρμες. Πρέπει να γίνει δημοκρατική συζήτηση για το εργαλείο αυτό και αυτό θα αποτελέσει και το κλειδί για να βρούμε την τελική ισορροπία στο θέμα. Πιστεύουμε ότι αν ε, ε, πετύχουμε να είμαστε διάφανοι, θα καταφέρουμε να δώσουμε μια απόκριση, θα παρακολουθήσουμε στενά τις απόψεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κυρία Κολπολανάτρη, και εγώ είμαι μηχανικός, δεν είμαι γιατρός. Ξεκίνησα την καριέρα μου με τηλεϊατρική για ένα νοσοκομείο παιδιατρικό στη Βοσνία. Και επειδή χρόνια δουλεύω στην υγεία, πρέπει να σας πω πως είναι η πρώτη φορά που θεωρώ πως τα ψηφιακά θα φέρουν τη διαφορά στις δυνατότητες θεραπεία των ασθενών και στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί ανεβαίνει το προσδίκημο ζωής, αλλά ε, δεν συνοδεύεται αντίστοιχα από αύξηση της ποιότητα αυτή τη αυτής της ηλικίας. 10 Απριλίου πολλά κράτη-μέλη ε, υπέγραψαν την ε, κοινή βάση δεδομένων για τα ιατρικά δεδομένα. Προσωπικά ιατρικά δεδομένα δεν θα υποσχεθούμε μόνο πιο ε, συγκεκριμένες παρεμβάσεις όταν έχουν προβλήματα οι πολίτες, αλλά και λιγότερο ακριβά, λιγότερο ακριβή ιατρική. Να τα πούμε με δύο λόγια και να ξαναδούμε την ψηφιακή κατάσταση, να σας στείλω ένα σημείωμα για όλα αυτά τα θέματα ε, στα οποία αναφερθήκατε. Χρειάζεται λοιπόν την ιδιαίτερη μας προσοχή. Αλλά αν υπάρχει κάποιος κλάδος όπου η δική μας ε, προσέγγιση θα φέρει διαφορά είναι αυτός. 36% όχι μόνο ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και οικονομική δραστηριότητα είναι το 6% του ΑΕΠ της Ευρώπης η ιατρική και είναι πάνω από το 10% της, ε, της δαπάνης ΑΕΠ ε, στα περισσότερα κράτη-μέλη και αυξάνεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο για τους δικούς μας πολίτες αλλά γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να ε, έχουμε σταθερά συστήματα πρόνοιας ε, στην Ευρώπη μέσω καινοτομίας και η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ε, και του big data στην ιατρική έχουν να κάνουν όχι μόνο με το πώς παραδίδουμε αυτά τα παραδοτέα, αλλά αν συγκριθούμε με την Κίνα και την ΕΠΑ και τις ΕΠΑ θα δείτε ότι εμείς την τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούμε σε καλύτερες τεχνολογίες υγείας και όχι στα καινούργια όπλα και ούτε στο να παρακολουθούμε ε, τις απόψεις κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, πολύ ενδιαφέρον και η εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών ε, κάνει την ε, ζωή μας πιο εύκολη. Έχουμε την ε, μεταφερσιμότητα των δεδομένων που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω πως δεν έχω χρόνο και θα αρχίσω να επιταχύνω. Όπως είπα λοιπόν και για τον κανονισμό θεωρούμε πως εδώ έχουμε ένα, κάνουμε μια αρχή που έχει ισορροπία, υπάρχει βέβαια όλη η διαδικασία συνομοθεσίας, είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεισφέρουμε και στη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, σαν αναφερθήκατε σε κάτι ε, πολύ σημαντικό που μιλήσατε στην πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες. Ελπίζω ότι από τις διαπραγματεύσεις που αυτή τη στιγμή γίνονται και είναι περίπλοκες ε, για τον κώδικα για τις καθολικές υπηρεσίες ε, θα μας βοηθήσει γιατί εκεί έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η μέση ταχύτητα ε, να εξασφαλίζεται παντού στην ε, εδαφική ε, στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Οπότε ελπίζω πως ο νέος κώδικας θα δώσει αυτές τις αποκρίσεις, θα επενδύσουμε περισσότερα ταμεία και όπου δεν έχει πετύχει τα αποτελέσματα αυτά η αγορά θα χρησιμοποιήσουμε με φυή τρόπο εθνικά και ε, τοπικά αλλά και ευρωπαϊκά ταμεία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ε, το Connecting Europe Facility με τα τρία δις θα κοιτάξει ακριβώς τις περιοχές όπου έχει αποτύχει η αγορά. Η συζήτηση μεταξύ προστασίας δεδομένων και ανοιχτών δεδομένων είναι μια συζήτηση η οποία θα παραμείνει ανοιχτή και ζωντανή. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μαγική λύση. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε τα ανοιχτά δεδομένα γιατί είναι το καύσιμο για πάρα πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη αλλά παράλληλα θέλουμε και ασφαλή δεδομένα και δεν θα έλεγα πως τα δύο βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Κάτι το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και εσείς το αναφέρατε είναι πως χρειάζονται περισσότερο ε, στην ε, αναγνωσιμότητα των δεδομένων και στο πού αποθηκεύονται και κυρίως να αποθηκεύονται στην Ευρώπη και θα δείτε πως το πρόγραμμα ψηφιακής Ευρώπης ένα μεγάλο κεφάλαιο θα έχει να κάνει με το θέμα αυτό, δηλαδή να μπορούμε εμείς να ανατρέχουμε και να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά στην Ευρώπη, κυρίως για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις στο ίδιο βάθος και όπως είπα είμαι έτοιμος να στείλω στη γραμματεία και μια, ένα σημείωμα με follow-up. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Γι' αυτό σας ζητήσαμε να έρθετε στην Επιτροπή. Διότι είναι κάτι που αφορά την κοινωνία μας στην Ευρώπη, αφορά το μέλλον της βιομηχανίας μας και άλλων τομέων όπως της υγείας. Πρέπει εμείς οι βουλευτές, όχι μόνο το κοινό, να γνωρίζουμε περισσότερα για αυτά που μέλλονται να, μέλλον να γίνουν. Ανεξάρτητα από το επάγγελμα, αν είναι κάποιος μηχανικός όπως εμείς, αν είναι γιατρός ή γνώστης θέματα τα φιλοσοφικά, να ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον και πώς θα καλύψει γρήγορο ίντερνετ όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για το μέλλον. Είναι σημαντικό για ιονδήποτε τομέα δραστηριοτήτων. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να σας ξανακαλέσουμε, ώστε να συζητήσουμε περαιτέρω αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε μεσημέρι, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ε, έχουμε συμμορφωθεί με το σχέδιό μας το χρονικό. Σπάνιο αυτό. Ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ενημερωθούμε τώρα για τις Η ε, κυρία για θέματα διακυβέρνησης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκροστέτ να σας πω ότι ο τρίτος τριμερής διάλογος έγινε στις 3 Μαΐου. Δεν είναι καινοφανείς οι πληροφορίες, είναι απειρχιωμένες, μπαγιάτικες και ο τέταρτο και ελπίζουμε τελικό τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για την 22 Μαου. Κυρία Γκροστέτ, ένα τρίλεπτο έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι, διεξήχθησαν τρει τριμερείς διάλογο 15 Μαρτίου, 10 Απριλίου και 3 Μαΐου. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι κάτι που περασπιστήκαμε στον τριμερή διάλογο. Με στηρίζουν οι δύο άλλοι συγητέ τη Επιτροπή Προπολογισμών και τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμήνη, είχαμε μία άποψη και προσπιστήκαμε τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Πολλά πολιτικά θέματα εξετάστηκαν πρώτα απ' όλα προπολογισμό. Ξεκινήσαμε από αντίθετε θέσει αρχικά όσον αφορά το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έκανε ένα βηματάκι στο δεύτερο τριμερή διάλογο. Πρότεινε 85% να διάταξη των ποσών. Εμείς προτείναμε 25% αλλά όπως θα καταλάβετε οι θέσεις ακόμα είναι πολύ μακριά και θέλουμε να αποφύγουμε στο μέγιστο δυνατό την αφαίρεση χρημάτων από υπάρχοντα προγράμματα. Όσον αφορά τους φορείς επιλεξίμους, χρειάζεται καλύτερη πλαισίωση των παρεκκλήσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τρίτες χώρες. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη εν μέρη τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου αλλά επενθυμίζω ότι είναι σημαντικό όλο τα άθρο για την επιλεξιμότητα να ενισχυθεί και όχι μοναδικά η παρέκκληση. Είναι ένα ουσιαστικό θέμα. Έχουμε ακόμα συζητήσεις από αυτού για το πρόγραμμα εργασιών. Συμβιβασμός πάντα συζητείται που θα επιτρέπει τη δικαιόλογηση της προσφυγής σε μια εκτελεστική πράξη. Το Κοινοβούλιο, υπενθυμίζω, ήταν υπέρ κατά πράξης. Θέλουμε να προσφυστούμε τα προνόμια του Κοινοβουλίου διευκρινίζοντας τον κανονισμό της κατηγορίες προγραμμάτων στις οποίες θα πρέπει να επισέθουν οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα. Ελπίζω ότι εκεί να καταλήξουμε χωρίς μεγάλες δυσκολίες σε μια συμφωνία. Οι δράσεις μη επιλέξιμες δράσεις Ακόμα επεξεργαζόμεθα το σχετικό κείμενο, το Συμβούλιο έχει κάποια προβλήματα να αποδεχτεί τη διατύπωση που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και εκεί πιστεύω ότι μια συμφωνία θα πρέπει γρήγορα να βρεθεί οι χρηματοπιστωτικές διατάξεις. Μπορέσαμε να πετύχουμε συμβιβασμό, δηλαδή να μην αναφέρουμε σε αυτά τα προγράμματα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά να προβλέπονται στο επόμενο πρόγραμμα μετά το 2020 που υπενθυμίζω ότι εκεί επεξεργαζόμαστε πρόγραμμα ένα 2019-2020 αλλά με την προοπτική συνεχίσεως των προγραμμάτων πέρα από το 2020. Για το πρόγραμμα 2009-2020 ουσιαστικά πρόκειται περί επιδοτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν. Εκεί βρήκαμε συμβιβασμό. Όσον αφορά τον, τον ελάχιστο αριθμό κρατών μελών, υπερασπιστήκαμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ελάχιστο αριθμό είναι τριών επιχειρήσεων που προέρχονται από τρία κράτη-μέλη για να δημιουργηθεί ένα ένα αντί δύο κράτη-μέλη που είχε προταθεί από το, Ευρωπαϊκό, από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο τελικά συμφώνησε με τη θέση μα, Μπορέσαμε να πετύχουμε συμβιβασμό που θα πρέπει να ικανοποιεί πολλού συναδέλφου του Κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά την δομή τη ε, της των πόνους, προσεγγίζουμε τη θέση των, του Συμβουλίου. Μπόνους χορηγούνται όταν ανήκει στον κατάλογο προγραμμάτων ΠΕΣΚΟ, τότε παίρνει μπόνους ένα πρόγραμμα, είτε όταν περιέχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όταν δίνει θέση στα mid ε, Εκφράσαμε την επιθυμία να έχουμε έναν μέγιστο άθισμα αυτών των πόνους, καθορίζεται στο 30% του κόστους του έργου αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να προβλέψουμε την χρήση των πόρων του προγράμματος και να επιτρέψουμε ένα μέγιστο, μέγιστη υποστήριξη προγραμμάτων, αριθμού προγραμμάτων. Συνόψισα, ξεπέρασα το χρόνο, ζητώ συγγνώμη, συνόψισα λοιπόν τα ουσιώδη των όσων πετύχαμε ή αυτών που συζητούνται. 22 Μαΐου είναι επόμενο τριμερή διάλογο. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια τελική συμφωνία εκεί. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχασε χρόνο, αλλά δυστυχώ Υπήρξε η απουσία της Κορεπέρ μεταξύ δύο τριμερών διαλόγων, μετά τα κράτη-μέλη τα οποία ε, δεν θέλουν, διστάζουν να προχωρήσουν. Ελπίζω λοιπόν την επόμενη φορά το Συμβούλιο να καταφθάσει με μια εντολή να διαπραγματευτεί και να καταλήξουμε σε κάποια ολοκλήρωση αυτών των συζητήσεων. Ευχαριστώ. Αξιέπαινο, ευχαριστώ πολύ, λέει ο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ε, πολύ περιεκτικές οι πληροφορίες λακωνικές περιγραφικές όμως. Βέβαια δεν είναι ο καλύτερος δυνατός ο χρονικός συντονισμός. Το θέμα της διακυβέρνησης είναι τώρα. Ο κ. Κροτούρμες θα μιλήσει για το governance. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα παραμείνω και εγώ στα γαλλικά. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται θα έλεγα με πολύ λογικό ρυθμό. Είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις και νομίζω πως είναι λίγο σαν να μαγειρεύει κανείς, θέλει να έχει κανείς και την κατάλληλη πίεση και την κατάλληλη θερμοκρασία και τα κατάλληλα συστατικά έτσι ώστε στο τέλος να φουσκώσει το κέικ και να είναι και εύπεπτο. Την τελευταία φορά κάναμε μια καλή συνταγή και καταφέραμε να απομπλοκάρουμε ένα θέμα το οποίο είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο ενέργεια, κλίμα και όλα αυτά εν ώψη του 2030 και νομίζω ότι εκεί τα πήγαμε καλά. Ε, βρήκαμε μια διατύπωση γιατί είπαμε πως εκεί στο παράρτημα θα δίδονται οι λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές. Αυτή ήταν μια καλή διατύπωση, έξυπνη διατύπωση και τους είπαμε εντάξει, ωραία, εσείς προετοιμάσετε ένα σχέδιο ε, και το σχέδιο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Πώς θα συγκρίνουμε τα σχέδια μεταξύ τους και η Προεδρία ε, τελικά παραδέχτηκε ότι η διατύπωση της δικής τους φρασιολογίας ήταν το λιγότερο ε, αμφίσιμη και θα δοθούν σχέδια για το 2030 με πάρα πολλές λεπτομέρειες και τα οποία θα είναι ολοκληρωμένα γιατί μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη έπρεπε να κάνουν σχέδιο για τις ΑΠΕ και μετά για την ενεργειακή απόδοση και μετά μια υποχρέωση για να κάνουν ε, σχέδιο για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και των δικτύων και αυτό που κάναμε μέσω της διακυβέρνησης είναι όλα αυτά τα σχέδια να είναι ολοκληρωμένα μέσα σε ένα σχέδιο κάτι το οποίο θα μας δώσει καλύτερη, γενικότερη άποψη και θα μου σε επιτρέψει να συγκρίνουμε για να δούμε ποιος κάνει τι και ίσως να κάνουμε ένα είδος διαγωνισμό των, με τους καλύτερους. Το άλλο σημείο στο οποίο προχωράμε είναι η πολιτική για το κλίμα. Εκεί έχουμε το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά και ένα σημείο πολύ σημαντικό είναι το μεθάνιο, γιατί σε επίπεδο διοξιδίου είμαστε 35-40% επάνω σε πομπές και η Καλιφόρνια εκτός από την πολιτική για το διοξίδιο του άνθρακα έχει και πολύ ε, στεναρή πολιτική για το μεθάνιο. Εκεί λοιπόν είπαμε σχέδιο για το μεθάνιο, αυτή είναι μια συμφωνία επί της αρχής και εκεί το μόνο που χρειάζεται είναι να δουλέψουμε λίγο τις λεπτομέρειες. Και ένα τρίτο σημείο που είναι θεσμικό είναι η πολιτική για το κλίμα, η οποία σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τους υπουργού ε, περιβάλλοντος και της ενέργειας στα χέρια των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας. Οπότε κάποια στιγμή είπαμε πως όλα αυτά θα πρέπει κάπως να τα συγκεράσουμε. Αλλά αν τα είχαμε κάνει, ε, θα είχαμε καταλήξει σε έναν μάλλον το χυλό, οπότε τώρα θα έχουμε δύο διαφορετικές επιτροπές και ό,τι είναι ε, καθαρά θέμα κλίματος θα μείνουν στους Υπουργούς ε, Κλίματος και ό,τι είναι καθαρά ενέργεια θα μείνει στα Υπουργεία Ενέργειας ή Οικονομικών και μετά προσπαθήσαμε, και αυτή είναι η βασική μας προσπάθεια, να δούμε ε, πώς μπορούμε αυτά να τα συνδυάσουμε. Θα γίνει και τριμερής διάλογος την επόμενη εβδομάδα, όπου ελπίζουμε να προχωρήσουμε για δύο θέματα. Ένα είναι η ενεργειακή ένδυα. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή δεν διαχειριστήκαμε καλά την κρίση των Lehman Brothers, έχουμε μια αύξηση των ε, φτωχών στην Ευρώπη και βέβαια η ενεργειακή ένδια και γιατί μιλάμε για ενεργειακή ένδια και όχι μεταφορική ή τηλεφωνική ένδια είναι ένα πραγματικό πρόβλημα σε πολλές από τις ανατολικές χώρες. Εκεί έχουμε και την κληρονομιά, αν θέλετε, των κτηρίων που είναι μάλλον σε κακή κατάσταση όπου μένει ο κόσμος σε ε, πολυκατοικίε οι οποίε είναι φτωχές, όχι πολύ ζεστές και δεν έχουν τα χρήματα για να τι ανακαινήσουν. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη που έχουν τέτοιου είδου προβλήματα για την ενεργειακή απόδοση να μπορέσουν να τα δουν όλα αυτά, να προχωρήσουν και το δεύτερο το οποίο θα προσπαθήσουμε αυτό είναι το τελευταίο που έχω να πω Euh, είναι το gap filler και να σε εξηγήσω τι είναι αυτό. Είναι ε, το υλικό με το οποίο γεμίζουμε τα κενά και έτσι μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα πρέπει να δούμε τι ποσοστό ΑΕ ε θα πιάσουν μέχρι το 2030 τα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν ένα πρώτο κενό. Εάν εμείς έχουμε ένα στόχο 35% ΑΠΕ, και τα κράτη-μέλη στις προτάσεις τους φτάνουν μόνο στο 33%. Έχουμε λοιπόν αυτό το κενό. Με ο ευρωπαϊκό στόχο 35 και κυβερνήσεις που στοχεύουν στο 33. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι να γεμίσουμε αυτό το κενό που θα είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε στα σχέδια τα για το, 320, για το 2030 με συγχωρείτε, να εξασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, ω στόχο τουλάχιστον, και αφού ξεκινήσει ο μηχανισμός θα πρέπει να παρακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη τροχιά, θα γίνει μια συζήτηση γραμμική, ενώ προτιμά μια καμπύλη η κυβέρνησή μας. Αλλά τουλάχιστον έτσι συλλογικά οι κυβερνήσεις το 21, το 22, το 23, το 25 μαζί θα επενδύσουν επαρκώ τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας έτσι ώστε να πετύχουμε τον ευρωπαϊκό στόχο ενώπιση του 2030. Αυτά είναι τα gap fillers, τα υλικά γεμίσματος ας πούμε. Και αυτά βέβαια αναλόγω με το τι θα γίνει στο Συμβούλιο και με την πίεση της Γαλλίας και Γερμανίας. Εμά η θέση μας είναι αυτή και ελπίζω πώς θα καταφέρουμε την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσουμε. Οπότε και θα γίνει ο τελευταίος τριμερής διάλογος τον Ιούνιο. Και βέβαια έχουμε δύο-τρία προβλήματα ακόμα να λύσουμε, αλλά έχω την ε, εντύπωση, γιατί εγώ είμαι πολύ έμπειρος μάγειρος, πως το έχουμε. Και μπορεί να τελειώσει το, το σχέδιο αυτό μέσα στην τρέχουσα προεδρία. Άλλη μια εύγλωτη παρουσίαση. Μέσα σε τρία λεπτά διαχειρίστηκες το χρόνο σου και τελείωσες. Στο μεταξύ όλα όσα είπες ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Euh, Μετά από το δεύτερο διάλογο νομίζω θα μπορέσουμε να έχουμε έναν τρίτο την επόμενη εβδομάδα και όλα αυτά θα, να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Τελευταίο θέμα, όχι όμως και ε, τελευταίο στο ενδιαφέρον, ε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το European Electronic Communications Code. Ε, είναι το... Η κυρία Καστίγιο ήταν πολύ... είχε μεγάλη υπομονή και θα την ρωτήσω τώρα να μας πει τι γίνεται με τον έκτο τριμερή διάλογο που έγινε στις 25 Απριλίου. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω τη μετρική μου γλώσσα για να είμαι πιο γρήγορη, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα μιλήσω λοιπόν πολύ γρήγορα και να σας πω πως κάθε φορά που εξηγώ πώς πάνε οι τριμερείς διάλογοι, έχω προσπαθήσει να σας ενημερώσω για το που πάει αυτή η νομοθετική πρόταση που έχει να κάνει με την αναθεώρηση τεσσάρων και όχι λιγότερο οδηγιών που ουσιαστικά αποτελούν αυτό το πακέτο το νομοθετικό που θα είναι η μελλοντική μας οδηγία. Είμαστε πια στην τελική φάση της διαδικασίας. Λέμε να τελειώνουμε τον Ιούνιο, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά. Και ο στόχος είναι να έχουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει κίνητρα για τις επενδύσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να έχει τις βέλτιστες δυνατότητες μετασχηματισμού ψηφιακού. Αυτή η επένδυση πρέπει να γίνει σε δίκτυα νέας γενιάς, έτσι ώστε να έχουμε σύνδεσιμότητα μέγιστη και νομίζουμε ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Χρειαζόμαστε 600 δις ή 500 δις ευρώ και θα πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό κλάδο γιατί εδώ και 10 χρόνια μιλάμε για αυτή την ανανέωση. Τελευταία φορά είχαμε το 2009 και έχουμε σκοπό να αναθεωρήσουμε και την προστασία των καταναλωτών και να διατηρήσουμε αυτή την αρχή του ανταγωνισμού και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου οι επενδύσεις στις υποδομές είτε στο φάσμα είτε στα δίκτυα να είναι πολύ ελκυστικό. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύνολο μέτρων. Υπέβαλε η Κομισιόν, συζήτησε το Κοινοβούλιο, έχουμε τη δική μας θέση και έχουμε μοιράσει σε δύο μεγάλους κλάδους την διαπραγμάτευση. Τρεις καλύτερα. έχουμε το κουτί της Πανδώρας, στο οποίο έχουμε βάλει όλα τα διάφορα θέματα που περισσεύουν και οι δύο μεγάλοι κλάδοι είναι το ραδιοελεκτρικό φάσμα και έχουμε ε, συμφωνία και έχουμε πολύ σημαντική πρόοδο, όπως ποτέ στο παρελθόν, για τη διαχείριση αυτού του φάσματος στα πλαίσια μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς και αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελική φάση της πρόσβασης στα δίκτυα νέας γενιάς. Και όλα αυτά είναι οριστικά για να δούμε τι είδους συνέπειες θα έχει αυτό σε επίπεδο του πόσο ελκυστικοί είμαστε για τις επενδύσεις. Και έχουμε και τον τελικό στόχο που είναι να έχουμε αυτά τα δίκτυα τα οποία θα είναι τόσο γρήγορα και τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού που χρειάζομαστε όλοι σήμερα. σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι στον επόμενο τριμερή διάλογο 22 Μαΐου αναφέρθηκε και η Φρανσουά στο θέμα αυτό, θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια συμφωνία για την πρόσβαση και θα περάσουμε στον τελικό που θα γίνει 5 Ιουνίου και αν όλα πάνε καλά, που είναι και η δική μας επιθυμία και των τριών ε, θεσμών, και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Κομισιόν θέλουν να τελειώνουμε και να σας δώσουμε την καλή είδηση που θα είναι πως ο φάκελος αυτός έκλεισε γιατί είναι ένα από τα πολλά πολύ σημαντικά κομμάτια της ε, νομοθεσίας μας και να φτάσουμε επιτέλους στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Και ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως αυτό το στοίχημα είναι τεράστιο και θα ήθελα όλα αυτά αναφέρουν το ποθητό αποτέλεσμα. Τα διαφούσα διακυβεύονται είναι τεράστια. So, thank you very much. We... Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το κλείσαμε το πρόγραμμα για σήμερα το πρωί. Τώρα το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε στις 2.30 με το σεμινάριο. Brexit και ενεργειακή πολιτική και εσείς και οι συνάδελφοι που λείπουν είστε καλοδεχούμενοι.